Okay, uh, we begin by the vote on the liability Να ξεκινήσουμε με την ψηφορία ευθύνη αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια. So, I understand you have your voting card. Έχετε έτοιμες τις κάρτες σας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στη συμβαστική 1. Ποιος είναι υπέρ. Against. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Είδα μόνο τέσσερα χέρια να σηκώνονται. Και πάλι υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε νομίζω ότι απορρίφθηκε συγγνώμη ηλεκτρονικά τη 44 παρακαλώ Όχι Ελέγχουμε τη 44 ηλεκτρονικά. We check 44. 44. Τη 44 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Περιμένουμε για την κυρία Ντελβό. reject. Απορρίπτεται σαφώς. 46 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ 48 Είστε υπέρ. Εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται δεν είδα όμως πολλά χέρια για να ελέγξουμε την 52 Adopted. 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 63 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Την 65. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Yeah. 66. 66 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά εποχέ. εγκρίνεται 16 υπέρ κατά εποχέ. εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται NV8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά εποχές να ελέγξουμε νομίζω ότι απορρίφθηκε 84 παρακαλώ εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ Συγγνώμη, είναι ταυτόσιμη. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Πάμε στη συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τοπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 6. 5. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φοβάμαι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές να ελέγξω παρακαλώ τη 14 εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά εποχές. Να ελέγξουμε και πάλι παρακαλώ. κρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 22 υπέρ κατά εποχές να ελέγξουμε 22 Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε, συγγνώμη εγκρίνεται και ένα υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε επίσης γιατί δεν είναι σαφές εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο της νομοδότησης ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Επομένως, συγχαρητήρια στον συγκεκριμένο που δεν είναι εδώ. application. Τώρα θα ψηφίσουμε την εφαρμογή της διαδικασίας Ευρώπης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής του κυρίου Χρυσόγονου. Okay. Uh, amendment 30 in favor. Against. Abstentions rejected. Uh, uh, 31 in favor. 31 υπέρ. Σας διακόπτω, αλλά εδώ δεν λειτουργούν οι, τα μηχανήματα ψηφοφορίας, οι συσκευές. Μπορείτε να μετακινηθείτε κάπου αλλού.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 κατά αποχές εγκρίνεται 52 αποσύρεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. αριθμό 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 Απορρίπτεται. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα πάλι με τις συσκευέ. Τα μάτια να λειτουργεί ξαφνικά. Ε, ψήφισα κατά, αλλά θα ήθελα απλώς να καταγραφεί. Ε, ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Συγχαρητήρια στον κύριο Χρυσόγωνο. Περάμε στην έκθεση Ντυρόν. Δηλώσει οικονομικών συμφερόντων των επιτρόπων. here. Συμβαστική βήτα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά Α, όχι, καταπίπτει. Πάμε στην 53. Ε, έχει αποσυρθεί ήδη. Αποσύρεται μάλλον. Κάπα. Τροσυμβαστική γάπα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Υπέρ κατά εποχές καταπίπτει Πεντεπτά καταπίπτει 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Hα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά απορρίπτεται ε, συμβαστική Α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 1, κοντ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 4 4-8 ε, υπέρ ε, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος ε, B, 4B, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4C, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4D, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 5, υπέρ, κατά,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 εγκρίνεται. 15α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σ υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επιβεβαίωση. D υπέρ, υιοθετήθηκε 15D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15E υπέρ κατά η ηλεκτρονική βεβαίωση πάλι. εγκρίνεται. 15F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15I υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 15J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται L ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15M υπέρ ο καταπίπτη 15N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15R υπέρ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 εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται παρόλο που δεν φαινόταν ότι θα εγκριθεί. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος α της αιτιολογικής έκθεσης υπέρ. Κατά. Αποχές. Πολύ λίγα χέρια. Επιβεβαιώνουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Παράγραφος β της αιτιολογικής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο της έκθεσης αυτή τη στιγμή. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Ντυρό. Now, the report of Uh, e Τώρα η έκθεση της κυρίας Κομοντίνη Κάτσια εν σχέση με μια συνεκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά ίσως να γίνει επαλήθευση. It's rejected. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται Έξι υπέρ κατά και πάλι θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Adopted. Εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό του ηλεκτρονικά. Χρειαζόμαστε. Λείπουν δύο ψήφοι. Could you move forward? Could you, Can you move to another seat, please? No, he hasn't got a card. Okay. Okay, okay. you're in favor. But you are in favor, I guess. Okay, so it's adopted. Γκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την κυρία Κομοντίνη. Και τώρα η έκθεσή μου για τη γενική αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού των, ε, του Κοινοβουλίου. prepared? Okay. So follow the chair voting. Λοιπόν. <laughs> Uh, amendment 7. Τροπολογία υπαριθμών 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3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 19. Είναι για τη διατύπωση. Υπέρ, κατά, 20. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 80 με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 συγγνώμη λέει ο πρόεδρος 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 71 επέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 επέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 επέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 επέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 επέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια στον εαυτό μου. Τώρα έχουμε τις μονομένες ψηφοφορίες. Καταρχήν έχουμε τον αριθμό 25. Θα το κάνουμε ηλεκτρονικά. That has been adopted. Εγκρίνεται. 27 και πάλι ηλεκτρονικά.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 Uh, dear colleagues, unfortunately, δυστυχώς να έχουμε καθυστερήσει κατά μισή ώρα. Ζητώ συγγνώμη καταρχήν από τον καθηγητή Φιλίπ Ντιπισού. Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ενρή Καπιτά. που θα μας παρουσιάσει τώρα το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κώδικα για το Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Επίσης θέλουμε να καλέσουμε τον κύριο Πορμπεζελόν, επιχειρηματία, τον Ντενίλα Σιρέρ, επίσης επιχειρηματία. Θα λάβετε τώρα το λόγο επειδή την προσκεκλημένη. Και θα ήθελα να μην μακρηγορήσετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιο χρόνο. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ ευγενικό να σας το ζητώ αυτό, αλλά παρόλα αυτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι της Επιτροπής, λέγομαι Φιλίπ Πισό, είμαι καθηγητής στο Παρί 1, Παντεών Σορβόνη και Γενικός Γραμματέας. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ, αν θέλετε να συνομιλήσετε, βγείτε από την αίθουσα. Είμαι Γενικός Γραμματέας ε, της Ένωσης Ερή Καπιτά, ε, η οποία έχει παρουσία σε 30 χώρες του κόσμου. Είμαι επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας μαζί με τον κύριο Μπός Βεσλούν, ο οποίος είναι εδώ και ήταν από τους εμπνευστέ ε, της οργάνωσης για την εναρμόνιση του δικαίου του επιχειρηματικού δικαίου στην Αφρική και θα θυμάστε υπήρξε ένα σχέδιο κώδικα για να υποστηριχθεί το επιχειρηματικό δίκαιο, το, δίκαιο των επιχειρήσεων στην Αφρική και είναι και ο Ντενής, ο οποίος εκπροσωπεί και την κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις. Ε, εδώ έχουμε την κοινωνία των πολιτών, ιδίως ο Πόρλ Μπεσλόν, ο ε, πέρσι εξέδωσε την υπόθεση ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο επιχειρήσεων δεν, θα, δεν μπορεί να είναι κατακαιρματισμένο ενώ η Ευρώπη έχει ένα ενιαίο νόμισμα τουλάχιστον τα 19 κράτη-μέλη. Έγινε υπόθεση ότι δεν θα μπορούσε να ευημερεί η Ευρώπη χωρί ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, δηλαδή να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες για τις επιχειρήσεις. Αυτό το έργο λοιπόν έγινε πριν το Brexit, αλλά... Μπροστά στο σεισμό του Brexit μπορούμε να αναρωτηθούμε αν ένα σχέδιο ευρωπαϊκού κώδικα δικαίου επιχειρήσεων ε, δεν θα μπορούσε να κάνει να αναβιωθεί το ευρωπαϊκό όνειρο και να δώσει όθηση στο ευρωπαϊκό κοδόμημα. Το έργο που έγινε από την Ενρή Καπιτό θα την παρουσιάσω εν συντομία. Πρόκειται για ένα έργο συνθετικής καταλαγοκοποίησης του κοινοτικού κεκτημένου σε 12 τομείς περιέργως ε, αυτή η δουλειά αξιολόγησης και καταλογοποίησης του κοινοτικού κεκτημένου, στο δίκαιο της αγοράς, στο δίκαιο ηλεκτρονικού εμπορίου, το δίκαιο εταιριών, το δίκαιο ασφαλίσεων, το δίκαιο εκτέλεση, το δίκαιο των επιχειρήσεων που είναι σε δυσκολία, το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο των ασφαλίσεων, το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησία, το φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο, διεξήχθη όλο αυτό το έργο σε συνεργασία με Ιταλούς και Γερμανούς νομικούς σε αυτούς τους 12 τομείς του δικαίου. Ποια είναι τα κύρια συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν αυτοί οι νομικοί. Σε αυτό το έργο, στο οποίο πρόλογο έχει γράψει ο πρόεδρος Βαλερίς Δισκάρντε Στέν, που έχει υποστηρίξει αυτό το έργο. Πρόκειται για ένα έργο που έχει επίσης μεταφραστεί σε γερμανικά και αγγλικά. Τα κύρια συμπεράσματα είναι τα εξής σε ό,τι αφορά τον τύπο υπερίσχυσε το συνέστημα ότι το δίκαιο των επιχειρήσεων ε, στην Ευρώπη υπέφερε από πρόβλημα προσβασιμότητας και κατανόησης, το οποίο συνδέεται με τον κατακαιρματισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωση και κρατών μελών και φυσικά με την αρχή της αναλογικότητας και της υπηκορικότητα. Αυτές οι αρχές αναλογικότητας και επικουρικότητας και ο κατακαιρματισμός ε, των αρμοδιοτήτων ήταν πραγματικά εμπόδια σε πραγματική ενοποίηση του δικαίου επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Και φτάνω στη δεύτερη παρατηρήσή μου που είναι Επί τη ουσίας, οι 14 νομικοί που εργάστηκαν επί αυτού του καταλόγου διεπίστωσαν δυστυχώ ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δίκαιου επιχειρήσεων 60 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης έμενε κάτι ανολοκλήρωτο σε μεγάλο βαθμό και ότι η δημιουργία ενός ενίου νομίσματος δεν συνοδεύεται από ένα δίκαιο επιχειρήσεων που είναι πραγματικά ομοιόμορφο. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο συχνά περιορίζεται σε θέματα που αφορούν κοινέ αρμοδιότητες μεταξύ Ένωσης και κρατών και το κοινοτικό κεκτημένο από όσο γνωρίζετε ε, βέβαια ε, αφορά και θέματα ανταγωνισμού που έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης οι συγγραφείς του καταλόγου εντυπωσιάστηκαν από κάποια τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενδιαφέρεται ή να νομοθετεί για ιδιαίτερες θεματικές, πάρα πολύ σημαντικές, όμως που έχουν ως στόχο να επανέρχονται ίσως υπερβολικά στην καρδιά της συζήτηση. Ε, θα αναφερθώ, παραδείγματο χάρη στην προληπτική εποπτεία των τραπεζών ε, και στην ε, εποπτεία της αγοράς, στα θέματα της διακυβέρνησης, εταιρικής διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της απάτης. Παρ' όλα αυτά, το συνέστημα που προέκυψε από αυτόν τον κατάλογο ότι αυτή η τάση της Ένωσης να επανέρχεται σε συγκεκριμένες θεματικές θα μπορούσε ε, ουσιαστικά να δώσει τροφή σε ευρωφοβικές θέσεις για ένα ευρωπαϊκό δίκαιο που θα είναι ουσιαστικά αποστεωμένο και είναι πιο χρηματοοικονομικό παρά εμπορικό. Με την ε, εξαίρεση των κανόνων για το ε, ηλεκτρονικό εμπόριο, την βιομηχανική ιδιοκτησία και τον ανταγωνισμό, αυτό το έργο μας επέτρεψε να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρεται τόσο για την καθημερινή πρακτική των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο γενικά έχουμε δύο πόλους που ήταν ε, στο επίκεντρο της συζήτησης του δικαίου των επιχειρήσεων, ο πόλος των χρηματοοικονομικών αγορών, των τραπεζών ε, και ε, Απ' την άλλη είχαμε το δίκαιο των καταναλωτών. Όμως ε, δεν ε, είδαμε να υπάρχει μια τέτοια ενοποίηση στο βαθμό που έχουμε ενιαίο νόμισμα. Έτσι λοιπόν μας εκπλήσει το εξής, το οικοδόμηση ενός δίκαιου εμπορικού ουσιαστικά υπολείπεται. Η υιοθέτηση του ενιαίου νομισματός δεν άλλαξε τα δεδομένα και αυτό μπορεί να φαίνεται κάπως παράδοξο. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε ουσιαστικά παρουσιάζονται κάποιες προοπτικές στον κατάλογο. Μία πρώτη προοπτική είναι να αναρωτηθούμε μήπως θα έπρεπε να ξαναθέσουμε σε εφαρμογή σημαντικά έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει από την Ένωση και από το Κοινοβούλιο. Παραδείγματο χάρη υπάρχει μια ιδιωτική ευρωπαϊκή εταιρεία. Επίση, του να υπάρχει ένα πραγματικό ευρωπαϊκό δίκαιο ε, συλλογική ε, αγωγής Επίσης, σκέφτομαι τη δυνατότητα να ε, φανταστούμε ότι θα έχουμε ε, ε, ευρωπαϊκές ασφάλειες και σκέφτομαι και το δίκαιο του ανταγωνισμού, το οποίο ουσιαστικά επικαλύπτεται. Νομίζω ότι κάθε μέρα γίνεται πιο παράδοξο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ένα νέο νόμισμα για τις εμπορικές του συναλλαγές, αλλά το δίκαιο των επιχειρήσεων να μένει εντελώς κατακαιρματισμένο, μάλλον σε μεγάλο βαθμό κατακαιρματισμένο. Και νομίζω ότι γίνεται όλο ένα και πιο αληθές, ότι η πλειονότητα των κρατών μελών έχουν ε, κοινό υπηρετικό δίκαιο και μπορούμε να φανταστούμε αν ένας κώδικας υπηρετικού δικαίου μήπως θα έπρεπε ε, ουσιαστικά να διαρθρώσει ε, την Ευρώπη των συναλλαγών για κάποιες ιδέες. Η πρώτη ιδέα, μήπως θα έπρεπε να κάνουμε πιο ευανάγνωστο το ευρωπαϊκό κοδόμημα στο δίκαιο των επιχειρήσεων, ενωποιώντα το σε έναν ευρωπαϊκό κώδικα δικαίου των επιχειρήσεων, το χάρη και να οργανώσουμε με διδακτικό και θεματικό τρόπο ουσιαστικά παίρνοντας τις οδηγίες ε, και τα νομοθετήματα στην τελευταία τους εκδοχή και ουσιαστικά να διευκολύνουμε με την ψηφιοποίηση και την μεταφορά στο εσωτερικό ιδέα λοιπόν ενός κώδικα δικαίου των επιχειρήσεων θα μπορούσε να το καθαστήσει πιο προσβάσιμο στους πολίτες και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να μπορούν να ξαναχρησιμοποιήσουν το δίκαιο της Ένωσης που δεν θα ήταν ένα δίκαιο που θα ερχόταν από αλλού. Και μακροπρόθεσμα είναι η δεύτερη υπόθεση που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να ενωρευτούμε, να αναρωτηθούμε μήπως θα έπρεπε ε, ε, νομίζω ότι μπορεί, έχει γίνει ήδη σε κάποιες ε, περιοχές στην Αφρική. Μήπως λοιπόν οι χώρες της Ένωσης να θεσπίσουν ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο του δικαίου των επιχειρήσεων για να προτείνουν και πάλι ένα πραγματικό κώδικα δικαίου των επιχειρήσεων που θα είναι ενοποιημένος και ομοιόμορφος και να αποτελεί το νομικό υπόβαθρο του ενιαίου νομίσματος που διέπει τις συναλλαγές εγώ θεωρώ, αλλά και οι συγγραφείς του καταλόγου, ότι γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο να συνεχίσουμε να κάνουμε εμπορικές συναλλαγές με ένα νέο νόμισμα, έχοντας διαφορετικά δίκαια. Γενικά, το νέο νόμισμα απαιτεί να έχουμε και νέο δίκαιο των επιχειρήσεων και δυστυχώς σήμερα ακόμη διακυβεύεται η οικοδόμηση ενό δικαίου επιχειρήσεων και νομίζω ότι αν είχαμε ένα κώδικα θα μπορούσε να αναβιώσει κατά κάποιο τρόπο και το ευρωπαϊκό όνειρο. Ευχαριστώ. Ε, Οι συναδελφοί σας που σας συνοδεύουν θέλουν να πάρουν το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που μας ε, καλέσατε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε σχέση με τα όσα είπε ο κ. Ε, ως κοινωνία των πολιτών να πω το εξή. Η κοινωνία των πολιτών μετά από τη χιλιοστή ευρωπαϊ... Ε, ελληνική κρίση του ευρώ τον Ιούλιο του 2015 αποφασίσαμε σύμφωνα και με παλιότερες ε, δεσμεύσεις που είχαμε στην Αφρικανική Ήπειρο με 250 εκατομμύρια ε, κατοίκους έχουν το ίδιο δίκαιο επιχειρήσεων εκεί. Αποφασίσαμε, λέω, να προσπαθήσουμε και υπογραμμίζω το προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών ε, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια ορμή, μια όθηση υπέρ της Ευρώπης. Ε, να σπρώξουμε την Ευρώπη υπέρ τη Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή οι πολίτε δεν ενδιαφέρονται πολύ για το μέλλον της Ευρώπης, δεν ξέρουν τι είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη όμω, ε, παρόλο που δείχνει απειρχιωμένο, είναι η ειρήνη για μα. Και η ειρήνη τι είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι, είναι το δίκαιο. Ξέρετε τι έκανε η Γερμανία. Το 1860 το πρώτο τούβλο της ε, γερμανικής ενοποίησης ε, είχε σχέση ακριβώς με την ενοποίηση του δικαίου των επιχειρήσεων. Η δική μας ε, αποστολή είναι να προσπαθήσουμε όλοι οι ακαδημαϊκοί, όλοι οι νέοι να συνεισφέρουν στη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού δικαίου. Ένα ενιαίο νόμισμα που δεν βασίζεται σε ένα ενιαίο κώδικα ε, ε, ε, δικαίου των επιχειρήσεων δεν μπορεί να σταθεί. Ο κ. Βαλερίδης Ζισκάρδεστα μαζί με τον Χέλμουντ Κόλ ξεκίνησε αυτό που έχουμε σήμερα και ο πρόεδρος Ζισκάρδεστα έλεγε χρειάζεται φορολογική ένωση για να στηρίξει την νομισματική ένωση. Ε, και, ε, και κάποιος... Ε, και, και, πρέπει να αναρωτηθούμε ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν φόρους, είναι αυτοί που εργάζονται, είναι οι επιχειρήσεις, ε, όλοι αυτοί δεν χρειάζονται τον ίδιο, να κινούνται στο ίδιο περιβάλλον σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε και κοινό δίκαιο των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να σας μεταφέρω τη μαρτυρία ενός ε, ε, επικεφαλής μιας μικρής ευρωπαϊκής επιχείρησης. Επισημένοντάς σας πόσο θα μπορούσε να αλλάξει η καθημερινότητα μιας μικρής επιχείρησης αν ο επιχειρηματής αυτός είχε μπροστά του και γύρω του ένα πιο πλατή πεδίο ε, από αυτό που έχει αυτή τη στιγμή. Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, δεν έχουν στρατούς δικηγόρων που να γνωρίζουν 19 διαφορετικά δίκαια. Και θα ήθελα να μπορούσα εγώ ως επιχειρηματίας να μπορούσα να αναπτύξω και να πουλήσω τα προϊόντα μου σε πιο πλατιά κλίμακα, κάτι που δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Προφανώς ε, αυτή η προσέγγιση δεν είναι προσέγγιση μιας μεγάλης ε, πολυεθνικής επιχείρησης που ε, έχει πρόσβαση σε άλλου τύπου κλίμακια. Τι όμως είναι η οικονομία. Η οικονομία μας, η ευρωπαϊκή οικονομία είναι το σύνολο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σκεφτείτε τις όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Σκεφτείτε όλες αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν ε, ένα ανοιχτό πεδίο, όχι στις 19 χώρες που έχουν δεχτεί το ευρώ μόνο. Φανταστείτε ε, να μπορούσε ο επιχειρηματίας αυτός να έχει πιο ανοιχτούς ορίζοντες απλώς. μια πρόσβαση, ανοιχτή πρόσβαση στις οικονομίες όλων των χωρών του ευρώ. Θα αύξανε πολύ την παραγωγή, τον κύκλο ε, ε, εργασιών, την απασχόληση και την ευημερία, τον πλούτο. Με αυτόν τον τρόπο θα ξανακατακτούσαμε την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Ιδεώδες. Οι νέοι συμμετέχουν μέσω του πρόγραμματος Εράσμους, αλλά <laughs> μετά όταν μπαίνουν στην πραγματική ε, οικονομική ζωή ε, απογοητεύονται. Θα ήθελα να συνεχίσουν να ονειρεύονται για την Ευρώπη και πιστεύω ότι μέσω του δικαίου, ξεκινώντας από το δίκαιο που αφορά την καθημερινότητα των επιχειρήσεων, που είναι αυτές που δημιουργούν τον ε, πλούτο και την ευημερία, θα ήταν ένας καλός τρόπος για να επανεφεύρουμε την Ευρώπη όπως λέει ο κ. Τιπισέ. Η οικονομική ανάπτυξη θα προεκυπτέ θα επέτρεπε, πιστεύω, να συγκλίνουν οι οικονομίες μας προς το κοινό νόμισμα. Γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το χάσμα είναι τεράστιο και όλο και πιο μεγάλο. Η, η, η ακριβής φύση του νέου, νομίσματος ακριβώς αυτό ε, μας επιβάλλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. πολύ κυρία για, για τις παρουσιάσεις σας αυτού του project. Πράγματι είναι πολύ εύλογα τα όσα λέτε. Και ακούγοντάς σας σκεφτόμουν τα λόγια του πρώτου Προέδρου της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλτερ Χάιν Χάουστάιν, ο οποίος έγραψε στο βιβλίο του ότι για πρώτη φορά η Ευρώπη ενοποιείται όχι μόνο μέσω βίας, πυρός και σιδήρου, αλλά μέσω μιας ε, πολιτιστικής ε, ισχύω που είναι το δίκαιο. Δεν ξέρω, έχουν οι βουλευτές ερωτήματα. Κυρία Χαουτάλα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις παρουσιάσεις. Χθες είχαμε μια πολύ, άλλη πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση εν σχέση με την σημασία της νομικής ε, ιστορίας όσον αφορά τα όρια και τις ε, δυνατότητες του ευρωπαϊκού οράματος. Ωστόσο, ποια είναι τα βασικά εμπόδια ε, σε σχέση με το πρίσμα ακριβώ της νομικής ιστορίας, ούτω ώστε να μεταβούμε προς έναν ενιαίο κώδικα επιχειρήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια οτοπία αυτό που προτείνουμε, αλλά είναι μια οτοπία που πραγματικά μπορεί να κάνει να πάλλονται οι καρδιές των Ευρωπαίων πολιτών, ξαναδίνοντας στην Ευρώπη ένα, ε, μια κανονιστική φύσεως φιλοδοξία η Ευρώπη έχει κληρονομήσει το ρωμαϊκό-γερμανικό δίκαιο και αυτό παρουσιάστηκε, αναπτύχθηκε πολύ καλά χθε. Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, εάν γίνει το Brexit, θα είναι χώρες αυτής ακριβώς της παράδοσης, η οποία κληρονόμησε την λογική της κωδικοποίησης των νόμων, οι οποίοι κωδικοποιούνται με έναν γενικό τρόπο και επιτρέπουν στους πολίτες να γνωρίζουν την εμβέλεια του νόμου και να συμμορφώνονται με τον νόμο. Ε, φαίνεται παράδοξο ωστόσο το ότι ένα ευρωπαίο νόμισμα δεν ανταποκρίνεται σε ένα ενιαίο δίκαιο επιχειρήσεων και είναι παράδοξο εφόσον πρόκειται για αν η Ευρώπη γίνει ε, ενωπηθεί όσον αφορά το υπηρετικό δίκαιο. Δεν υπάρχει ένα δίκαιο των επιχειρήσεων, γιατί ακριβώς είναι ένα δίκαιο των επιχειρηματικών συναλλαγών. Το γεγονός ότι έχουμε δεχθεί μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο μοντέλο πρόσληψης του δικαίου, γιατί το δίκαιο πραγματικά ε, είναι, φέρει, διατυπώνει συγκεκριμένες αξίες. Είναι στοιχείο πολιτιστικό, είναι στοιχείο ρύθμισης μιας χώρας και είναι ένα στοιχείο που σχετίζεται με την ακτινοβολία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει σαν αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μπορούν να βιώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι σαν μια τροχοπέδη, όχι σαν ένα καταναγκασμό και όχι όπως λένε οι ευρωσκεπτικιστές ε, ε ακριβώς ότι είναι, έχει μια καταναγκαστική φύση η Ευρώπη. Αντίθετα, υπάρχει μια ενότητα μεταξύ των επιχειρήσεων. Συζητώντα με Γερμανού συναδέλφου ή, Γερμανού, ή Ιταλούς συναδέλφους, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφορές που όμω μπορούν ε, πολύ καλά να, να γίνουν αντικείμενο επεξεργασία και κωδικοποίηση. Αυτό έγινε στην ε, Μαύρη Αφρική, όπου κανείς, όπως ξέρετε, δεν ε, προχωράει σε συναλλαγές χωρίς να ε, ε, απευθύνεται στο δίκαιο το οποίο ισχύει που αφορά τις πιστώσεις, τη φύση των συναλλαγών κλπ. Και ξέρουμε ότι, στην, ε, ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό αυτό. υπάρχουν δύο άλλοι ομιλητές, θα πρέπει παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οργανισμό Αρή Καπιτάν που ήρθε ιδιαίτερο στο συνάδελφό μου, καθηγητή κύριο Ντεπισό. Και θεωρώ ότι η άποψή του είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρουσα γιατί μας παρουσίασε ότι το γεγονό ότι υπάρχει ένα νέο νόμισμα θα συνεπάγεται ένα ενιαίο κώδικα του δικαίου των επιχειρήσεων. Ε, είναι απολύτω θεμητή αυτή η προοπτική και εκτιμώ τον ενθουσιασμό με τον οποίο ο κύριος Ντοπισό ε, υπερασπίστηκε την άποψή του. Εγώ απλώς ε, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν και άλλες ε, απόψεις γιατί είμαι αυτό που ο κύριος Ντοπισό ονομάζει ευρωσκεπτικιστή. εγώ θέλω να μια παρατήρηση απλώς. Δεν έχει πολεμικό χαρακτήρα η, τα όσα θα πω. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί πιστεύουν όλο και μια ε, μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ε, θεωρώ ότι η εκείνος πιστεύει ότι εγώ θεωρώ ότι το, το αφρικανικό μοντέλο ίσως ε, ταιριάζει για τους Αφρικανούς μεν, αλλά όχι για τους Ευρωπαίους. Και όταν ο κύριος καθηγητής λέει ότι ίσως θα γίνει το Brexit, εγώ πραγματικά σοκάρομαι να ακούω αυτά, διότι ήδη αποφάσισε ο Βρετανικός λαός και ε, θα πρέπει να το σεβαστούμε. Και πραγματικά δεν είναι αυτό το όραμα των Ευρωπαίων. Έχουμε ε, λίγο χρόνο. Κύριε Ντουράν, θα είμαι πολύ γρήγορος γιατί μπορώ να απαντήσω στον κύριο Τεμπρετόν. Ε, κύριε Ντουπισό, ε, ο πατέρας σας νομίζω ήταν πρίτανης του Πανεπιστημίου στο οποίο σπούδασα στο εμπορικό δίκαιο και το εταιρικό δίκαιο. Άρα συμφωνούμε, είμαστε στην κοινή γραμμή. Τώρα θέλω να πω στον κύριο Ντεμπρετόν, είσαστε νομικός και εγώ το ίδιο. Θέλετε να μου εξηγήσετε πώς ε, θα μπορούσε να συγκροθεί το γαλλικό δίκαιο χωρί το ρωμαϊκό δίκαιο και μπορείτε να μου εξηγήσετε τι θα ήταν η δημοκρατία χωρί την ιστορία τη Ελλάδα στην Ευρώπη. Υπάρχει μια στιγμή όπου η βούληση να θέλει κανεί. Ε, που θα πρέπει κανεί να απευθυνθεί, να παραπέμψει στην ιστορία του δικαίου. Και εσεί ε, γνωρίζετε ότι πόσο σημαντική είναι η ιστορία του δικαίου. Γιατί δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το παρόν εάν δεν στραφούμε στο παρελθόν. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην εγγραφούμε σε μία. Να μην εγγράψουμε το παρόν σε μια ιστορική προοπτική, γιατί είναι το παρελθόν αυτό το οποίο επέτρεψε την έλευση της δημοκρατίας και την πρόοδο του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη είναι εξή. Ε, μ' αρέσει ο ενθουσιασμό μου, γιατί ε, και το όραμα της Ευρώπης ε, πραγματικά το συμμερίστηκα στην, ε, στο παρελθόν με τον Κον Θα ήθελα να πω το εξή. Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στο σωστό χώρο για να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Γαλλία, εκείνη και άλλα ευρωπαϊκά κράτη δεν ε, προασπίζονται αυτή την ε, λογική της Ευρώπης και η Γαλλία συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών των χωρών. Η Γαλλία βλέπει τις Βρυξέλλες και την Ευρώπη σαν ένα πεδίο μάχης. Λέμε ότι πιστέψαμε ότι τις Βρυξέλλες με μία νίκη. Δεν πρόκειται για μία κοινή βούληση ολοκλήρωση της Ευρώπης. Αν θέλετε, πρόκειται για ένα πεδίο μαχών. Αυτό το οποίο θέλετε θεωρώ ότι μπλοκάρετε από κάποιες λογικές, εθνικιστικές, κρατιστικές και περιορισμένες. Δυστυχώς... Δεν έχουμε χρόνο, ζητώ συγγνώμη, λέει ο κ. Ε, δυστυχώς... Ε, ο κύριος Λεμπρετών μιλάει για κυριαρχία, τώρα δεν ξέρω αν μιλάει για την κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ε, κρατών εθνών. Ε, θέλετε και εσείς το λόγο. Ο κύριος Ντουρό πήρε τα, τις λέξεις από το στόμα. Εμείς ε, πουλάμε σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν έχουν όλοι οι αγοραστές μας τα ίδια δικαιώματα. Ε, και εγώ είμαι μέλος της ε, κοινωνίας των πολιτών και βλέπω ότι υπάρχει μια στρέβλωση ε, ανάμεσα ε, στον συνάδελφο που είναι και αυτός καθηγητής και σε μας. Εγώ καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας. Δεν είναι δυνατόν να πουλήσει κανείς ένα κόσμημα σε έναν Άγγλο και να σου, μπορεί να σου το επιστρέψει ε, ενώ το γαλλικό, σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο η, η αγοροπολισία έχει ολοκληρωθεί. Ε, παλιότερα ε, που πληρώναμε με τσεκ σε ευρώ και μας λέγανε ότι αυτό δεν είναι νόμισμα παλιότερα λέω, οι Γερμανοί το κάνουν αυτό Χρειάζονται επίσης ε, ρύθμιση και στις συλλογικές αγωγές. Οι συλλογικές αγωγές θα πρέπει να είναι παντού ίδιες. Είτε κανείς είναι κυριαρχικός, είτε όχι, ε, είτε είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό στο δυτικό κόσμο, έτσι, είμαστε στο δυτικό κόσμο, αυτό μην το ξεχνάμε. Entre Νομίζω ότι ο κόμπο είναι στο ότι πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στο ρωμαϊκό και το βρετανικό αγγλοσαξονικό δίκτυο. Νομίζω ότι οι φιλοξενούμενοι μας ε, ε συμμετείχαν σε μια παθιασμένη συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση ειλικρινή. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή. Δεν είχαμε για πολύ χρόνο σήμερα. Θα φροντίσουμε να μην ήταν αυτή η τελευταία φορά που μιλήσαμε για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί ομιλητές, αγαπητοί συμμετέχοντες, ε, ξεκινάμε την ακρόαση για τις προοπτικές του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου για την εκδίωξη των εγκλημάτων του Ισλαμικού κράτους εναντίον γυναικών και κοριτσιών ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που οργανώνεται από κοινού με την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Αυτή τη φορά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ακρόαση γιατί συνδέεται με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που έχει σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα συζητήσουμε το θέμα της λογοδοσίας ε, για τα εγκλήματα που διαπράχθησαν από το αποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος ε, του Ιράκ και του Αλσάμ, της ευρύτερη Συρίας, που είναι γνωστό και ως Άϊσις. Κατά μάχων και κατά μειονοτήτων στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Πριν να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποια αντίρρηση γιατί βρίσκεται εδώ η τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πάλι TV και βιντεοσκοπή. Λοιπόν, καθώς ε, θα συζητήσουμε για τη δίωξη εγκλημάτων ε, κατά κοριτσιών και γυναικών και θεωρήθηκε ότι είναι σωστό για το λόγο αυτό να συνδιοργανώσουμε με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συγγνώμη, με των γυναικών. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Βεζάκο Μέντα Λόπε, ε, που είναι αντιπρόεδρο στην Επιτροπή ΦΕΜ και ευχαριστώ για την με βοηθάτε να συμπροεδρεύσουμε. Επίσης, η ακρόση αυτή αφορά θέματα για τα οποία είναι αρμοδίες οι επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΝΤΡΟΑ. Και οι πρόεδροι των δύο αυτών επιτροπών έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στην ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση, ελπίζω, που θα ακολουθήσει τις παρεμβάσεις των ομιλητών. Και τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω στην ακρόση μας την αντιπροσωπεία ε, της ε, μειοψηφίας για ζήτη, της μειονότητας για ζήτη, με συγχωρείτε, που προέρχεται από την περιοχή Σιντζάρ και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωσή μας. Καλώς ορίσατε. Χωρίς χρονοτριβή, θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Ζώπη Μέντα Λόπες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως ε, υπόθηκε, είμαι και εγώ εδώ για να δώσουμε το σήμα έναρξη σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ μετά στις επιτροπές μου για αυτή τη συνεργασία. Δεν ε, είναι τωρινή, έχουμε συνεργαστεί και με άλλες επιτροπές και επίσης ε, θέματα σχετικά με αυτό που θα συζητήσουμε και σήμερα. Θυμάμαι μια κοινή ακρόαση που οργανώθηκε με τις Επιτροπές Σέντε και Ντρουά πέρσι για την κατάσταση των γυναικών σε εμπόλεμες ζώνες. Και πιστεύω φυσικά ότι πρόκειται για ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σκόπιμο χρονικά, καθώς βλέπουμε ένα πλαίσιο ε, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική που αφορά τον εξτρεμισμό, ένα πλαίσιο εξτρεμισμού και δεν αφορά μόνο το Ισλαμικό κράτος, τον ΤΕΣ, αλλά και άλλες ριζοσπαστικές ε, ακραίες μάλλον δυνάμεις όπως είναι η Αλνούσρα και η Αλκάιντα. Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το διεθνές πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται η Ευρώπη και έχουμε συζητήσει το τελευταίο έτος το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης και των προσφύγων. Έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες και μεγάλη περιέργεια να ακούσω τις παρεμβάσεις των προσκεκλημένων. Έχω μία πολύ μεγάλη περιέργεια για το πώς ε, ουσιαστικά θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα εγκλήματα κατά γυναικών και κοριτσιών, κατά γυναικών και παιδιών, αλλά να δούμε και το θέμα των αιτιών. Δηλαδή, πώς δυνάμει του διεθνούς δικαίου θα καταπολεμήσουμε τις αιτίες δημιουργίας αυτών των ακραίων δυνάμεων και του εξτρεμισμού και μάλιστα πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε και το φαινόμενο της χρηματοδότησης αυτών των οργανώσεων. Δεν θα χρονοτριβήσω περαιτέρω. Θα ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για να περάσουμε στην ακρόαση. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, κύριο Ζερόμ Τέντιν, ο οποίος ε, είναι ερευνητής στην Ακαδημία της Ιρέης για το ανθρωπιστικό δίκαιο, δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικό δίκαιο. Έχει εργαστεί ο προσκεκλημένος μας και ως ε, νομικός στο ειδικό δικαστήριο για το Λίβανο. Θα έχετε το λόγο για τα επόμενα 15 λεπτά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ε, πρόσκληση. Δυστυχώς παίρνω το λόγο με λύπη γιατί έχουν ε, γίνει κάποιες, ε, κάποια εγκλήματα κυρίως κατά γυναικών και κοριτσιών κυρίως στην Μέση Ανατολή αλλά και στη Βόρεια Αφρική όπου βασιλεύει το Ισλαμικό κράτος. Απογοήτευση, επειδή η Ευρώπη και η διεθνή κοιμότητα δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια συνεκτική και αποτελεσματική στρατηγική για να θέσουν τέλος αυτή τη βαρβαρότητα και για να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές συνέπειες. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζω την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα για να συνεισφέρει στο να θέσει σε εφαρμογή δικαστικές λύσει προκειμένου να ξεριζώσουν αυτή τη βία και να ανακουφίσουν αυτούς που υποφέρουν, τις γυναίκες και τα παιδιά. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω το θεσμικό περιβάλλον στο οποίο τέτοιες λύσεις θα έπρεπε να τεθούν σε εφαρμογή σε διεθνές επίπεδο. Θα αφήσω στους υπόλοιπους ομιλητές ε, ε, τη δυνατότητα να αναφερθούν λεπτομερώς ε, στις δυσκολίες της προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών σε εμπόλεμε καταστάσεις. Και θα ξεκινήσω με δύο θέματα που θεμήθηκα όταν γνωστοποίησατε το θέμα. Καταρχήν, γιατί η δίωξη των εγκλημάτων του ISIS θα έπρεπε να αφορά κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά κατά προτεραιότητα. Ε, ε, ουσιαστικά δρά αυτή η οργάνωση κατά όλων των ατόμων που δεν συμφωνούν με την ιδεολογία της ε, χωρίς ε, να λαμβάνει υπόψη το φίλο την ηλικία, τη θρησκεία. Ε, ουσιαστικά έχουμε δει χριστιανούς, μουσουλμάνους, γεζίδι να στοχεύονται και πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση είναι θεμελιώδης για την προστασία γυναικών και κοριτσιών γιατί τονίζει τη σοβαρότητα βίων πράξεων που συχνά αγνοούνται και το, γεν... το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι οι άνθρωποι αυτοί, δεν λαμβάνεται παρκώς υπόψη από το διεθνές ε, σύστημα. Ακόμη και αν έχει γίνει πρόοδος ε, σε αυτό το τομέα από την ε, τότε που η αναγνώριση των Διεθνών Ποινικών Δικαστηρίων για την πρώην Ιουκοσλαβία και τη Ρουάντα αναγνώρισαν ότι οι σεξουαλικές πράξεις, οι πράξεις σεξουαλικής βίας μπορούν να αποτελούν εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Συγγνώμη, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά για τη διερμηνία. Επίση, σε κάθε προσπάθεια δικαιοσύνη που έχει ληφθεί σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου τι ακόλουθε πέντε προτεραιότητε, Καταρχήν, να ποινικοποιηθούν όλε οι μορφέ βία και σεξουαλική βία ε, που ε, γίνονται κατά αυτών των κατηγοριών ανθρώπων. Δεύτερον, να θεσπίσουμε πολιτικέ έρευνε και ποινική δίωξη και να θετήσουμε κανόνες ε, διαδικασίας και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που να είναι κατάλληλε. Τρίτον, να προβλέψουμε τα μέτρα προστασίας και ψυχολογικής υποστήριξης ε, που χρειάζεται η ακρόση των θυμάτων. Τέταρτον, να βρούμε μορφές αποζημίωση που να λαμβάνουν απόψη την ιδιαιτερότητα αυτών των βιοπράξεων και να προσλάβουμε τέλος κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να υποστηρίξει και να προστατεύσει τα άτομα αυτά. Το δεύτερο θέμα ε, το οποίο ξέτασα ήταν ε, να δω γιατί ενδιαφέρεστε μόνο για το Ισλαμικό κράτος. Πραγματι, υπάρχουν και άλλες ε, τρομοκρατικές ομάδες, η Αλκάιδα, η Αλνόσρα, η Μπόκο Χάραμ, καθώς ε, και ε, οι δυνάμεις του Συριακού καθεστώς επίσης προβαίνουν σε μαζικά εγκλήματα, εγκλήματα τα οποία αν μείνουν ατιμόρυτα, πραγματικά δεν θα υπάρξει καμία προσπάθεια συμφωλίωσης και πρέπει να δεκτώ ότι κυρίως δίνεται μία έμφαση στον ΤΕΣ και στα εγκλήματα που διαπράττει. Τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας φαίνεται όλοι να είναι στο ίδιο μήκο κύματο σε σχέση με την αναγκαιότητα να ενώσουν τις δυνάμει τους για να μειώσουν, για να νικήσουν, να αποδυναμώσουν αυτή την οργάνωση που θεωρούν ομόφωνα τρομοκρατική. Υπάρχει και το ψήφισμα 2244 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 20 Νοεμβρίου 2015 που ομόφωνα, μέσω του οποίου το Συμβούλιο ζητά συντονισμό δράσης από τα κράτη-μέλη προκειμένου να θέσουν τάλους στις τρομοκρατικές ενέργειες του ISIS και να εξαλείψουν ε, αυτό το ιερό που έχει δημιουργήσει στο Ιράκ και στη Συρία. Σίγουρα θα πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να ε, αποδείξουν ε, ότι δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα ε, ουσιαστικά δρούν όπως ε, ξέρουμε, με κάποιες πολιτικές που συχνά είναι αδιαφανείς και ε, πολλές ε, φορές αγνοούν πολλές άλλες καταστάσεις και πολιτικούς ή στρατιωτικούς ηγέτες που θα έπρεπε να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Έτσι, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε και το, το δικαστικό, διεθνές δικαστικό σύστημα λειτουργεί ατελώς. Θα πρέπει να γίνει καλύτερα όμω μια προσπάθεια, ακόμη και αν είναι τελής, παρά να μην γίνει τίποτα. επίση. να υπογραμμίσω ότι τόσο ο διεθνικός χαρακτήρας ορισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων όπω το ISIS, όπω και η απειλή που θέτουν στο σύνολο των κρατών απαιτούν μια συντονισμένη δικαστική δράση σε διεθνέ επίπεδο. Αυτέ οι δύο προηγούμενε παρατηρήσει, κατόπιν αυτών των δύο προηγούμενων παρατηρήσεων, ερχόμαστε τώρα στο επίκεντρο του θέματο. Η διεθνής κοινότητα ε, τι μπορεί να κάνει σε δικαστικό επίπεδο για να καταπολεμήσει αποτελεσματικά και τα εγκλήματα που διαπράττουν από το ISIS κατά γυναικών και κοριτσιών. Θα ξεκινήσω από την εξή διαπίστωση. Οι διεθνεί δικαιοδοσίε συχνά δεν μπορούν να δράσουν με μεροληψία και ανεξαρτησία σε συνθήκε πολέμου που πλήττουν ε, τα εδάφη που είναι τώρα κυρίω ε, υπό τον έλεγχο του ISIS στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία ή στην Ιεμένη. Στο πλαίσιο αυτό, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο φαίνεται ως η ιδανική λύση φυσικά. Ασκεί μια σχεδόν παγκόσμια ευθύνη και μόνιμη και μπορεί να ενεργοποιηθεί κάθε στιγμή από το Συμβούλιο Ασφαλείας όταν υπάρξει απειλή στην ειρήνη και στην παγκόσμια ασφάλεια η κατάσταση στην οποία βρίσκεται φυσικά, βρίσκονται τα κράτη, ε, αποτελούν μια τέτοια απειλή. Λιβύη, η Συρία, η Εμένη επίσης. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια και φυσικά έχει την απαραίτητη υποδομή και ε, το καθεστώς του μπορεί να του επιτρέψει να ε, θεωρήσει τα σεξουαλικά εγκλήματα ως εγκλήματα πολέμου και μιλάμε για διάφορες μορφές βίας όπως είναι ε, η σεξουαλική υποδούλωση, η εξεργαστική πορνεία, ο βιασμός ε, κτλ. Έχουν ε, προσληφθεί και εμπειρογνώμενες το 2014 το γραφείο του Εισαγγελέα δημιούργησε και μια πολιτική που αφορούσε τα σεξουαλικά εγκλήματα και την εισαγωγή διακρίσεων φύλου προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή την αρχή της συμπληρωματικότητας προκειμένου να παρουσιαστούν αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο. Όλα φαίνεται ότι αρκεί να καλέσουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να διώξει και να δικάσει όσους διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα από το ISIS. Όμως υπάρχουν τρία μεγάλα εμπόδια για αυτές τις λύσεις σε πολιτικό, θεσμικό και νομικό επίπεδο που, μπορούν, που μας οδηγούν να σκεφτούμε άλλες λύσεις. Σας δούμε συντομία αυτά καταρχήν σε πολιτικό επίπεδο. Γνωρίζετε ότι η αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου ασκείται σε σχέση με μια κατάσταση και καταλαβαίνουμε ε, τι λέει το άρθρο 13 του κανονισμού του. Χωρίς να μπούμε στις λεπτομέρειες, θα πρέπει να πούμε ότι ορίζεται από κάποιες γεωγραφικές ε, παραμέτρους. Δηλαδή όλη την επικράτεια μιας χώρας εντός της οποίας έχουν διαπραχθεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ε, ή γενεκτονίες. Άρα, Κανένα κράτος, ωστόσο ε, το Ισλαμικό κράτος δεν ε, έχει επικυρώσει αυτό το κανονισμό. Ε, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα έπρεπε να αποφασίσει να αποθύλει ατομικά ατομικές προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο στη βάση αποφάσεων που έχουν ληφθεί βάσει του άρθρου 4 του, της Διεθνούς Χάρτας. Ε, το να βρεθεί μια συνένεση αυτό δεν είναι πιθανό. Και αυτό θέτει το ευαίσθητο θέμα ε, της δίωξης στο Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί από μια διασυνεργική οργάνωση, δηλαδή μια οργάνωση ε, τη δευτερότητα της οποίας επεκτείνεται σε πολλές χώρες. Σε θεσμικό πλαίσιο γνωρίζουμε ότι το δικαστήριο πραγματικά είναι υπερφορτωμένο από υποθέσεις που αφορούν πολλές ε, χώρες, την ακτή Ελεφανταστού, τη Γεωργία, τη Λιβύη, το Μαλί, την Ουγκάντα κλπ. Το Κονγκό και το Σουδάν. Ε, και για να δώσουμε μόνο ένα αριθμό, το Διεθνές Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία χρειάστηκε 20 χρόνια για να ολοκληρώσει το, έργο του, ενώ ε, εξέταζε μια σχετικά απλή υπόθεση, δηλαδή μια χώρα, την πρώην Ιουγκοσλαβία. Άρα, ε, τι μπορούμε να περιμένουμε από το Διεθνές ε, Δικαστήριο. Θα ήταν ε, λογικό να επιφορτήσει το δικαστήριο αυτό με το επιπρόσθετο έργο να διώξει τα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπραχτεί από, το, από την ΤΑΕΣ σε πολλές χώρες και μάλιστα και σε πολλές υπήρους. Ίσως θα χρειαζόταν να αναθεωρηθεί το σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να μετατοπιστούν οι δραστηριότητε του σε όργανα τα οποία να συσταθούν στι εν λόγω χώρες. Και θα έπρεπε στο δικαστήριο αυτό να... Εάν δίδονταν στο δικαστήριο αυτό περισσότερε αρμοδιότητε, θεωρώ ότι αυτή η στρατηγική θα ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Ε, βεβαίως δεν μπορώ να αρνηθώ τι προσπάθειες που γίνονται εκ μέρους του δικαστηρίου για να εγγραφεί η αρμοδιότητά του, ε, να ισχύσει η αρμοδιότητά του σε ορισμένες ε, υποθέσεις. Ωστόσο, το έργο αυτό δεν θα είναι πολύ εύκολο να εκπληρωθεί σε σχέση με τρομοκρατικέ ομάδες, των οποίων η ιεραρχία δεν είναι πολύ κατανοητή, διάκριτη δεν αρνούμε την προσπάθεια που κάνει το δικαστήριο και να δικάσει αποτελεσματικά εγκλήματα τα οποία εμπίπτουν στην δική της αρμοδιότητα. Ωστόσο, δυστυχώς, όποια και αν είναι εμβέλεια αυτών των προσπαθειών, δεν θα μπορέσει ποτέ να ε, εκπληρώσει αυτό το πρόκληση, να αντιμετωπίσει την πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει. Μία τρίτη δυσκολία νομική φύσεω θα πρέπει επίση να αναφερθεί. Μία οργάνωση σαν την Daesh κάνει τρομοκρατικέ δραστηριότητε που χαρακτηρίζονται ω εγκλήματα πολέμου εφόσον διαπράττονται στο πλαίσιο μια ένοπλη σύραξη ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εφόσον γίνονται στο πλαίσιο μιας μαζικής και συστηματικής επίθεσης κατά του άμαχου πληθυσμού αλλά επίσης διαπράκτη, διαπράττει τρομοκρατικές ε, πράξεις σε κατάσταση ειρήνης, εκτός αυτού του πλαισίου πολέμου, όπως για παράδειγμα στο Βέλγιο, στη Γαλλία ή στο Λίβανο. Έτσι λοιπόν, ε, τα εγκλήματα αυτά δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Ε, σε ορισμένε χώρες τα εγκλήματα αυτά μπορούν να εκδικαστούν από την εθνική δικαιοδοσία, σε άλλες όχι. Θα ήταν λοιπόν ευκταίων αυτές οι... Ωστόσο θα ήταν ευκταίο αυτές οι τρομοκρατικές πράξεις να μην παραμείνουν ατιμόρυτες. Και θα πρέπει για αυτές να ισχύσει η διεθνής ε, δικαιοδοσία. Η... Ε, ε, και συνεπώς η λύση θα ήταν ίσως η σύσταση ενός διεθνούς δικαστηρίου ad hoc. Ε, στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει ίσως να εξετάσουμε τη σύσταση ενός δικαστηρίου από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η αρμοδιότητά του θα πρέπει να επεκτείνεται σε όλα τα εδάφη στα οποία δραστηριοποιείται το ΝΤΑΕΣ, το Ιράκ και στη Συρία και να περιλαμβάνει όλα τα εγκλήματα τα οποία έχει διαπράξει αυτή η οργάνωση συμπεριλαμβανόμενων και των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά γυναικών και παιδιών καθώς και ε, καθαρά τρομοκρατικέ ε, πράξεις. Θα πρέπει να έχει μια διασυνορική διάσταση, θα πρέπει να έχει όλα τα ανακριτικά μέσα και τα μέσα να επιληφθεί ποινικά αυτών των υποθέσεων ε, και να συμπεριλαμβάνει βεβαίω και τα σεξουαλικά εγκλήματα. Λαμβάνοντα υπόψη την εμπειρία των ad hoc δικαστηρίων, η αποτελεσματικότητά του θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά συγκεκριμένα εάν οριστούν κάποιοι δικαστές ανακριτές ε, και το κόστος των δικαστηρίων θα μπορούσε να είναι πολύ μειωμένο σε σχέση με τα, το κόστος, τα έξοδα των διεθνών δικαστηρίων. Ε, γιατί στην περίπτωση αυτών των προσωρινών δικαστηρίων οι δικαστές ε, ορίζονται κατά περίπτωση και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εγώ είχα, ε, ε ήμουν υπάλληλο στο ειδικό δικαστήριο για το Λίβανο που ήταν ε, πρωτοπόρο όσον αφορά την απόδοση διεθνούς δικαιοσύνης για πολλά χρόνια και είχε ακριβώς την πρωτοβουλία να προετοιμάσει το κανονισμό ενός μόνιμου δικαστηρίου που να επιδικάζει τρομοκρατικές υποθέσεις. Ε, την εποχή εκείνη ε, δεν είχε δοθεί μεγάλη προσοχή στο καθεστώς και στον κανονισμό αυτού του δικαστηρίου ε, γιατί οι χώρες μέλη δεν είχαν ιδιαίτερη διάθεση να ασχοληθούν με τον τομέα αυτό. Αλλά θεωρώ ότι σήμερα θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα βάση εργασίας στην περίπτωση που τα, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα να προωθήσουν μια δικαστική πρωτοβουλία για να καταπολεμήσουν την ΝΤΑΕΣ και τις άλλες θερμοκρατικές οργανώσεις. Ελπίζω με την ομιλία μου να σας έδωσα κάποια ερίσματα για να συζητήσετε την αντιμετώπιση εγκλημάτων κλιμάτων της ΝΤΑΕΣ και άλλων οργανώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα λάβει το λόγο η δόκτωρ Κρίστεν Κάμπελ από το Goldsmith College. Το κολέγιο Goldsmith είναι βασική ερευνήτρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, ε, το οποίο έχει ένα χρηματοδοτούμενο ε, ε, πρόγραμμα τετραετές ε, για την ε, δίωξη ε, των εγκλημάτων φύλου. Εξετάζει την, τέτοιες διώξεις ενώπιον του ε, Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Ιουγκοσλαβία και την Βοσνία. Ε, Δόκτωρ Κάμπελ, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρόγραμμα μας, το ερευνητικό μας πρόγραμμα εστιάζεται και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Ιουγκοσλαβία, πρώην Ιουγκοσλαβία και στο θέμα ε, το, και, και, στο θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα. Ε, δύο διδάγματα από τις ε, διώξεις εγκλημάτων, σεξουαλικών εγκλημάτων ε, στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Η, ανάγκη πρώτον καλών βέλτιστων πρακτικών και δεύτερον τη σημασία του να συνδέσουμε την ε, διολογοδοσία σε διεθνές επίπεδο μαζί με τις διαδικασίες, δικαστικές διαδικασίες μετά την, το τέλος των συγκρούσεων. Δεν μιλώ για συμφιλίωση έτσι. Ε, ας δούμε ποιες είναι οι βασικές ε, προκλήσεις, τα βασικά προβλήματα που έχουμε σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές. Ε, Αυτά τα προβλήματα έχουν σχέση με τα εξής πέντε. Πρώτον, πρώτο πρόβλημα είναι η χρήση ε, ερευνητικών διαδικασιών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Το δίδαγμα εδώ πέρα από το Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία ήταν ότι παρόλο ότι ε, η, Επιτροπή που ερεύνησε τα πρώτα, καταρχήν τα γεγονότα, είχε περιορισμένο εύρος και βεληνικέ, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το έργο τη για τι κατοπινές διώξει. Η ενδεχόμενη σημασία και ο περιορισμός των ερευνητικών διαδικασιών και από τη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας και οι πιο περιορισμένες ε, έρευνες σε ε, κάθε δικαιωτικά όργανα θα πρέπει να λεφτούν υπόψη διότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τις διώξεις αργότερα. Δεύτερο πρόβλημα, ε, δεύτερη πρόκληση, ε, είναι θέματα που έχουν σχέση με τα πιστήρια αλλά και με το ουσιαστικό δίκαιο. Ε, το ουσιαστικό δίκαιο αφορά περιορισμό του πεδίου αυτή τη στιγμή διότι υπάρχει εθιμικό δίκαιο το οποίο διεθνές και ε, ε, εθνικό εθνικό δίκαιο το οποίο περιορίζει πάρα πολύ ε, την, το πεδίο του ουσιαστικού δικαίου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, ε, υπάρχουν κενά στα, στο νομοθετικό πλαίσιο και πεδία ασάφειας τα οποία δημιουργούν προβλήματα Ας πάρουμε για παράδειγμα τα, ε, τα ουσιαστικά σημαντικά, τα, κέρια ε, αδικήματα, γενοκτονία για παράδειγμα. Ε, υπό το εθνικό δίκαιο δεν προβλέπεται προστασία. Ε, οι γιαζίδοι ας πούμε δεν υπόκεινται σε προστασία και όμως θα πρέπει να προστατευτούν. Επίσης, ε, στο, τα δικαιώματα κατά ε, τα, τα δικαιώματα της ανθρωπότητας προβλέπουν ε, ορισμένου τέτοιου τύπου αδικήματα. Ε, δεν είναι σαφές ότι περιλαμβάνουν τις γυναίκες ως ξεχωριστή ομάδα. Τέλος, έχουμε και ε, εγκλήματα πολέμου το ερώτημα όμω είναι αν αυτοί οι κανόνες που αφορούν τα εγκλήματα πολέμου έχουν γενική ισχύ, αν έχουν δηλαδή διεθνή χαρακτήρα. Επίσης, στην πράξη υπάρχει και το θέμα της ε, συσταλτικής ή περιοριστικής εφαρμογής των κανόνων για τα πιστήρια. Πολύ συχνά έχουμε δει ανακρίσεις και έρευνες ε, που εφαρμόζουν με διαφορετικό τρόπο τα κριτήρια. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα παρανόησης ε, της νομικής ε, ευθύνης. Για παράδειγμα, το πώς είναι δυνατόν να καθοριστεί ποιος ήταν ο επικεφαλής. Επίσης έχουμε και προβληματική εφαρμογή κανόνων για πιστήρια, όπως πολύ συχνά ε, ζητούνται υψηλής ποιότητας πιστήρια, ε, για να ε, ε, αποδειχθούν αδικήματα από εφιστάμενους. Συνήθως αυτά θα πρέπει να τέτοιου είδους ποιότητα θα πρέπει να αφορά τους επικεφαλείς. Τρίτον, θα πρέπει να εντοπιστούν επαναλαμβανόμενα αδικήματα και ο χαρακτήρας τους. Για παράδειγμα, διαφορετική τύπη σεξουαλικής βίας σε τέτοιου τύπου ε, συγκρούσεις. Ε, είναι δύσκολο να συνδέσουμε τη σεξουαλική βία που συνδέεται με μια ε, σύγκρουση με άλλου τύπου αδικήματα που έχουν σχέση με το φύλλο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε στο περιβάλλον τους τα αδικήματα αυτά σε, όπου λαμβάνουν χώρα και άλλου είδους άνομες και παράνομες πράξεις. Χωρίς αυτή την προσέγγιση Δηλαδή χωρίς να εντοπίσουμε τα επαναλαμβανόμενα αδικήματα είναι δύσκολο να χαρακτηρίσουμε σωστά τα αδικήματα και να διώξουμε όλους τους τύπους της σεξουαλικής βίας και της βίας κατά του φίλου. Θα πρέπει να κάνουμε τη σύνδεση ανάμεσα στους ε, αυτούργους και στις ομάδες στις οποίες ε, ε, ανήκουν. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος, ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι θύματα, όπως επίσης και άλλες ομάδες αυτούργων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε ποιες είναι οι κοινότητες και οι ομάδες που έχουν πιο πολύ ε, πληγή από τέτοιου είδους αδικήματα. Δεν είναι δηλαδή πρόβλημα να εντοπίσουμε τη δράση μα στι συγκεκριμένε ομάδες. Τέταρτον, στερεότυπα για το φύλλο και παρανοήσει. Και εδώ πάλι αυτό σχετίζεται με όλες τις πτυχές ε, των, διεθνών και εθνικών συστημάτων. Τέτοιου τύπου παρανοήσει είναι, για παράδειγμα, ότι η σεξουαλική βία αποτελεί διεθνέ αδικήμα μόνο αν αποτελεί αντικείμενο πολιτική ή στρατηγική ή μιας ε, ε, θεώρηση ότι ε, τα θύματα αρνούνται να καταθέσουν εξαιτία του στιγματισμού. Ε, το Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία έδειξε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα σωστό. αυτά αποτελούν κοινωνικά στερεότυπα, αλλά το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς διώξεις δεν θα πρέπει να αναπαράγουν αυτά τα στερεότυπα. Τέλος, μπορούμε να μιλήσουμε και για θεσμικά εμπόδια. Και αυτό το έχει σχέση με εμπόδια και στο επίπεδο της ανάκρισης και στο επίπεδο της δικαιοδοσίας. Ε, για παράδειγμα, ίσως δεν υπάρχουν επαρκείς γνώσεις και προσόντα, επαρκείς τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά τις διώξεις αυτές, ε, έλλειψη αποφασιστικότητας και βούλησης ε, ή αδυναμία εφαρμογής πολιτικών ε, σε όλους τους τομείς του δικαιοδοτικού συστήματος. Υπάρχει και ένα άλλο και μια άλλη ομάδα προβλημάτων που έχουν σχέση με την διεθνή ποινική λογοδοσία και τις διαδικασίες που θα λαμβάνουν χώρα μετά το τέλος των συγκρούσεων. Η διεθνής ε, ποινική ε, λογοδοσία ε, θα πρέπει να ενταχθεί στους συνολικούς στόχους. Πρέπει να συνδέσουμε την διεθνή ποινική λογοδοσία με τις ευρύτερες ε, δικαστικές διαδικασίες στο τέλος των συγκρούσεων, έτσι ώστε να μην ξανασυμβούν αυτά τα αδικήματα. Η δίωξη σεξουαλικής βίας και αδικημάτων ε, φύλου στο δικαστήριο της πρώην Ιγκολαβίας απέδειξε ότι πρέπει να συνδέσουμε τη διεθνή, τις πρωτοβουλίες διεθνούς ε, ε, ε απόδοσης δικαιοσύνης με τις, με τις συνολικές διαδικασίες, νομ, δικαστικές διαδικασίες. Διότι οι διεθνείς διαδικασίες δεν μπορούν ποτέ να διώξουν όλους τους ε, αυτούργους παρά μόνο μερικούς από αυτούς. Ε, αυτή είναι η φύση της διεθνούς ε, ποινική διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να λάβουν, ε, και οι εθνικές δικαιοδοσίες. Επίσης, διώξεις θα πρέπει να ενταχθούν στις διαδικασίες, δικαστικές διαδικασίες μετά το τέλος της, των συγκρούσεων. Για παράδειγμα το Διεθνές Δικαστήριο την πρώην Ιγκοσλαβία πολύ συχνά κατηγορήθηκε ότι δεν συνέδεσε τις δραστηριότητε του με περιφερειακά και εθνικά δικαστήρια. Αυτό άλλαξε και η αλλαγή αυτή ήταν πολύ σημαντική για να συνεισφέρει στις ε, διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μετά το τέλος της σύγκρουσης στην πρώην Ιγκοσλαβία. Τέλος, αν πούμε ότι θέλουμε να διώξουμε αυτά τα εγκλήματα, τότε θα πρέπει να συμπεριλάβουμε πολιτικές γυναικών και φίλους σε αυτές τις ε, διαδικασίες. Γιατί χωρίς αυτό θα έχουμε πολιτικές οι οποίες χειρίζονται ότι προσφύγουν τα συμφέροντα των θυμάτων, αλλά δεν θα το κάνουν. Μόνο με αυτή την προσέγγιση μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των διεθνών συστημάτων δικαιοδοσίας. Ε, ε και, ε, γιατί ε, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να παρασπιστούμε τα συμφέροντα των θυμάτων. Αυτές οι διώξεις θα πρέπει να γίνονται σε επαφή με τα θύματα και τις οργανώσεις τους. Η κατακαιρματισμένη προσέγγιση ε, των αδικημάτων αυτών, για παράδειγμα, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, ε, ήταν ε, ε, ιδιαίτερα προβληματική για τα θύματα. Ένα σημαντικό σημείο είναι πώς μπορούν να ενταχθούν αυτές οι στρατηγικές στη λογοδοσία. Πρέπει διεθνή στάνταρ διώξεων, διεθνείς προδιαγραφές ε, ε, να ενταχθούν στις εθνικές δικαιοδοτικές διαδικασίες και θα πρέπει να έχουμε μηχανισμούς ε, εφαρμογής και παρακολούθησης. Επίσης, χρειάζεται να έχουμε προδιαγραφές ποινική και αστικής λογοδοσίας σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζονται συγκεκριμένες στρατηγικές για ποινικέ διώξεις σε εθνικό και, διεθνε, και διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, αποζημιώσεις, ε, ψυχοκοινωνική υποστήριξη κλπ. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια διτή στρατηγική για την διεθνή ποινική λογοδοσία. Αφενός θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα επαρκές νομικό πλαίσιο για τις ε, διώξεις με βάση βέλτιστες πρακτικές και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, ένα σύνολο από ε, αρχές για τις μετασυγκρουσιακές διαδικασίες που θα συμπεριλαμβάνουν εθνική, ποινική και αστική λογοδοσία. Αυτό είναι τεράστιο έργο. Και πριν τελειώσω θέλω να υπογραμμίσω Ποιε είναι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας για να προκειμένου να ακολουθήσουμε αυτή τη διτή στρατηγική. Οποιοδήποτε νέο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να, ε, προσεγγίζει τα εξής επτά σημεία. Και αυτά είναι τα πιο βασικά σημεία, εντάξει. Πρώτον, η ανάπτυξη ε, στοιχείων εγκρήματος, ε, τρό, τύπων νομικής ευθύνη και προδιαγραφών για τα πιστήρια. Δεύτερον, θα πρέπει οι διώξει να γίνονται μέσα σε, στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο είναι τα αδικήμενα, τα αδικήματα. θα πρέπει να εντοπιστούν συγκεκριμένα, συγκεκριμένοι τύποι πράξεων και δράσεων που αποτελούν αδικήματα. Ένα άλλο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι η ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη για μάρτυρες που είναι είτε αρσενικού είτε θηλυκού φύλου. Το δεύτερο κομμάτι αυτής της στρατηγικής είναι οι αρχές πλαίσιο, το πλαίσιο αρχών για την μετασυγκρουσιακή εποχή. Πρέπει οι γυναίκες να συμπεριληφθούν και να συμμετάσχουν ενεργά ε, καθώς ε, στις διαδικασίες αυτές, καθώς επίσης να ενταχθούν και πολιτικές για το φύλλο ε, αυτές, σε αυτές τις διαδικασίες. Μόνο έτσι μπορούν να πετύχουν. Δεύτερον, Πρέπει να αξιολογήσουμε το κενό ε, που υπάρχει, τα κενά που υπάρχουν ε, σε εθνικό επίπεδο στην ε, αστικές και ποινικέ διαδικασίες σε σχέση με, τα, με, το, με τις αντίστοιχες διεθνείς διαδικασίες. Τρίτον, θα πρέπει να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τις διώξεις. Πώς ξέρουμε αν είναι αποτελεσματικές οι διώξεις αυτές. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν καλύπτουν όλα τα θύματα ε, και όλους τους θύτες. Τέλος, η πρόβλεψη αποζημιώσεων οικονομικής στήριξης, ε, ψυχοκοινωνικής στήριξης κλπ. είναι απόλυτα σημαντικά στοιχεία έτσι ώστε πραγματικά να αγγίξουμε όλη την κοινωνία. Χωρίς αυτή τη διετή στρατηγική, αυτό που, μένει είναι απλώς μια διεθνής ε, δίωξη από μόνη της, απομονωμένη, με συχνά φτωχά αποτελέσματα. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβασή σας. Τώρα θα ήθελα να καλέσω τον, κύριο, τον καθηγητή Σεντρικ Ρένχαρτ από το Πνευματισμό της Ουτρέχτης να πάρει το λόγο και να σχολιάσει το θέμα της λογοδοσίας μη κρατικών παραγόντων από τη σκοπιά του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Και πάλι έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. κ. Δεντίν επικεντρώθηκε στο θέμα τη λογοδοσία από τα διεθνή ποινικά δικαστήρια και η Δ. Κάμπελ ω ένα βαθμό. Επίση, εγώ τώρα θα αναφερθώ σε, κάποια, σε κάποιους λογοδοσία, μηχανισμούς λογοδοσίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε την ε, κυρία στοιχεία τη παρουσίασή μου σήμερα. Θα αναφερθώ στο θέμα τη ποινική λογοδοσίας στα εθνικά ε, δικαστήρια και κυρίως στα δικαστήρια των κρατών μελών καθώς ενδιαφέρεστε περισσότερο για αυτά και κατόπιν θα αναφερθώ στο θέμα της αποζημίωσης και της αγωγή αποζημίωση για ηθική βλάβη σε εθνικά δικαστήρια και πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση το θέμα των διοικητικών κυρώσεων κατά των υποστηρικτών του ISIS και τέλος, αν έχω χρόνο, το θέμα της κρατικής ευθύνης, γιατί και τα κράτη ίσως να είναι ή συνυπεύθυνα για τη διάπραξη ε, αυτών των πράξεων βίας. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι για την πρώτη βουλά εδώ. Ε, βλέπετε ε, το αν δεσμεύονται οι ένοπλες ομάδες ε, από το δίκαιο του πολέμου και φυσικά είναι σκόπιμη αυτή η ερώτηση καθώς το ISIS είναι ένοπλη ομάδα και θα πω κάτι που θα αποδεικνύει ότι δεσμεύεται από αυτό το δίκαιο. Η πρώτη ερώτηση, οι ένοπλες ομάδες δεσμεύονται από τον νόμο. Ναι, είναι η απάντηση. Αναμφισβήτητα, το άρθρο 3 της Σύμβασης της Κοινωνίας επιβάλλει ε, κάποιες υποχρεώσεις σε κυβερνητικούς αλλά και με κυβερνητικούς ε, παράγοντες. Αυτό υπάρχει και στο Διεθνές Εθνικό Δίκαιο, όπως μας επιθυμεί η Διεθνής Επιτροπή του Ρυθμού Σταυρού το 2005. Τα κράτη και οι ομάδες δεσμεύονται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ε, προκειμένου να δρουν υπό ίσους κανόνες. Διαφορετικά μόνο οι κυβερνήσεις θα δεσμεύονταν στο πεδίο της μάχης. Είναι σαφές λοιπόν ότι παραβιάζει το ISIS, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, όταν διαπράττει σεξουαλικά εγκλήματα όμως το θέμα είναι το θέμα της συγκατάθεσης. Νομικά κανένας δεν έχει συγκατατεθεί στο να δεσμεύεται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Δεν είναι κράτος, άρα δεν ανήκει στις συμβάσεις της γυναίκες. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να σχεστεί κανείς ότι οι κανόνες της Σύμβασης της Γενέβης αλλά και στο Διεθνές Εθνικό Δίκαιο μπορεί να μην είναι νόμιμες γιατί ε, βλέπετε ε, ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ για την ομιμότητα των κανόνων, το πώς αντιλαμβανόμαστε την ομιμότητα. Τώρα, ε, ουσιαστικά μία λύση μπορεί να είναι να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τη συγκατέθεση. Φυσικά, μία ΜΚΟ στην Γενέβη που λέγεται Τζενίβα Κόλ προσπαθεί να, να υπογράψουν αυτές ε, οι μη κρατικέ οργανώσεις σε κάποιες πράξεις δέσμευσης έτσι ώστε να δεσμεύονται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Υπάρχει μια πράξη για τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών και Τζενίβα Κόλλη επίση δραστηριοποιείται στη Συρία και έχει ουσιαστικά αποκτήσει μια δέσμευση από τι ε, κουρδικέ δυνάμει αυτοάμυνα ε, που ξέρετε ότι έχουν και μάχη με ομάδε γυναικών. Επίση η Τζενίβα Κόλ συνομιλεί με άλλε ομάδε, όμω μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει να διασφαλίσει αυτέ τι πράξει δέσμευση. Όμω δεν συνομιλεί με το ISIS. Όταν συζητούμε για θέματα συμμόρφωσης για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δικαίωμα θα πρέπει να πείσουμε τις ε, ένοπλες ομάδες ότι οι αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου δεν ε, αφορούν μόνο τον νόμο αλλά υπάρχουν και στο δικό τους πολιτισμό. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το 2009 οι Ταλιμπάν ε, από όλες τις οργανώσεις προώθησαν το δικό τους κώδικα ε, δεοντολογίας για την συμμόρφωση με το νόμο του πολέμου. Τώρα βέβαια είναι διαφορετικό όταν σέβονται το διεθνές δικαίωμα, υπάρχουν κάποια ανοίγματα. Να προσθέσουμε όμως ότι υπάρχει ένας νομικός κίνδυνος όταν συνομιλεί κανείς με τις ε, ένοπλες ομάδες. Υπάρχει ένας ε, κίνδυνος ε, δίωξης και στο κράτος σου όταν το χάρη συνομιλείς με αυτούς μπορεί να σε καταδικάσουν ότι μπορεί να υποστηρίζεις τους τρομοκράτες. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που ουσιαστικά πρέπει να επισημάνουμε ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μπορούσε απευθυνθεί στο κράτος για αυτά τα θέματα. Τώρα, Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια για την ε, λογοδοσία. Ήδη ακούσαμε ότι τα δικαστήρια στην περιφέρεια μπορεί να μην είναι τα κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν, να δικάσουν αυτά τα εγκλήματα. Θα μπορούσαμε όμως να θεσπίσουμε, να ιδρύσουμε ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο ή να παραπευθούν οι άνθρωποι αυτοί ήδη σε ένα υπάρχον δικαστήριο. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι κάθε κράτος ε, έχει το δικό του ποινικό δίκαιο και ίδιο και στην Ευρώπη και ε, υπάρχει και στη Συρία ένα κέντρο δικαιοσύνης και λογοδοσίας ε, σε μια πρόσφατη έκθεσή του είπε ότι αυτή είναι η πιο βιώσιμη επιλογή λογοδοσίας ε, βραχυπρόθεσμα πριν ε, να δημιουργηθεί ένα διεθνέ ποινικό δικαστήριο. Έχουμε αυτά τα δικαστήρια ούτω ή άλλω. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν ποινικά δικαστήρια που μπορούν να ασκήσουν δικαιοδοσία και σε δικού του υπήκοου αλλά και σε υπήκοου τρίτων κρατών υπό την αρχή τη παγκοσμία δικαιοδοσία. Σε ό,τι αφορά την αρχή της ε, εθνικότητας. Ξέρουμε ότι έχουμε κάποιους επικόους κρατών μελών που πολεμούν στην περιοχή και αυτοί ε, σίγουρα έχουν διαπράξει τέτοια εγκλήματα. Ένα αριθμός λοιπόν υποθέσεων ε, έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια. Κάναμε μία έρευνα στην Τρέκτη, όμως σχετίζονται οι υποθέσεις αυτές με υποστήριξη των τρομοκρατών, με δολοφονίες, αλλά όχι με σεξουαλικά εγκλήματα αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα ε, η κυρία Κάμπελ. Έτσι λοιπόν, ίσω να χρειαστεί να αλλάξουμε νοοτροπία. Επίση, ε, μπορούν να ασκήσουν τα δικαστήρια παγκόσμια δικαιοδοσία. Δεν χρειάζεται ε, σύνδεσμος. Απλώς αυτό έχει να κάνει με τη σοβαρότητα του εγκλήματο και κανεί δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η σεξουαλική βία είναι ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα. Τώρα, συχνά, τα κράτη, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα απαιτούσαν την εδαφική παρουσία του παραβάτη. Περισσότεροι από αυτού του παραβάτε φυσικά δεν είναι εδώ, παραμένουν στην περιοχή. Τεχνικά λοιπόν δεν υπάρχει δικαιοδοσία. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι από αυτού τους δράστες έχουν φύγει στο εξωτερικό και έχουν έρθει στην Ευρώπη και ε, ακούσαμε και μία αναφορά στο έχουμε μαζική έλευση ανθρώπων από τη Συρία. Κάποιοι μπορεί να είναι βέβαια υπό παρακολούθηση, αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν ακόμη ζητήσει και άσυλο. Κάποιες ε, μεταναστευτικές αρχές ίσως ε, θα έπρεπε να δώσουν την απαραίτητη προσοχή, θα έπρεπε να ε, αρνηθούν την αναγνώριση βάσει του άρθρου 1F της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχει σύνδεση με τους εισαγγελίες. Η καλύτερη ε, πρακτική είναι στην περίπτωση Γερμανίας το 2015 οι μεταναστευτικές αρχές έδωσαν πάνω από 2.000 φακέλους ε, ανθρώπων που τους υποπτεύονταν ότι έχουν διαπράξει εγκλήματα στη Συρία και στο Ιράκ και αυξήθηκαν οι διώξεις. Δεν έχουμε όμως ακόμη καταδίκες για περιπτώσεις σεξουαλικών εγκλημάτων και δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες όπως και να έχει, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να απευθυνθεί στις αρχές μετανάστευσης για να ενισχυθεί η συνεργασία και να θέσουν ως προτεραιότητα το θέμα της δίωξης ε, δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων. Ένα δύσκολο θέμα είναι η συλλογή αποδείξεων. Ξέρουμε ότι οι ανακριτές δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη Συρία ε, για να κάνουν έρευνα στην ίδια τη Συρία. Εξαρτώμαστε λοιπόν σε μάρτυρες εκτός της Συρίας ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν λάβει συνεντεύξεις. Επίσης μπορούμε να βασιστούμε στον έλεγχο των κινητών και σε ε, διαδικασίες ε, εξέτασης ασύλου. Ε, έχουν υπάρξει κάποιοι μάρτυρες που έχουν κληθεί να μιλήσουν και υπάρχει συνεργασία μεταξύ ανακριτών και θα μπορούσε να ενισχυθεί. Επίσης, θα ήθελα να αφήσω στην προσοχή σας το γεγονός ότι τα Ενωμένα Έθνη πρόσφατα υπόγραψε μια συμφωνία με την Αραβική Λίγκα προς αυτή την κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση. Η κύρια πρόκληση σας είναι να πείσουμε τα θύματα να εμφανιστούν. Όμω ε, ίσως η κυρία Κάμπελ αναφερθεί, εγώ δεν είμαι ειδικό στη σεξουαλική βία. Κατόπιν, περνάμε στι αγωγέ αποζημίωση για ηθική βλάβη στα εγχώρια δικαστήρια. Εδώ δεν μιλώ για τεχνική λογοδοσία, αλλά για την αποζημίωση που θα δοθεί στα θύματα. Ξέρουμε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο υπάρχει και δυνατότητα να ζητήσει κανείς αποζημίωση, αλλά εδώ αναφερούμε σε διαδικασίες ενώπιον των εγχώριων διαδικαστηρίων, ε, και των ε, δικαστηρίων χωρών που βρίσκονται ε, γύρω. Τα θύματα μπορούν να κάνουν μία προσφυγή ακόμη και αν δεν κάνει κάτι ο εισαγγελέα. Μπορούν τα θύματα να πάνε και σε ένα αστικό δικαστήριο, όμω υπάρχουν προβλήματα, ότι υπάρχει σύνδεσμο με την Ευρώπη. Μπορούν όμω να υπερβληθούν αυτά τα νομικά προβλήματα. Υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν διάταξη που λέγεται ε, το Δικαστήριο Αναγκαιότητα, Forum of Necessity, δηλαδή κατά εξαίρεση μπορεί να δικάσει το δικαστήριο προκειμένου να μην υπάρχει άρνηση απονομή δικαιοσύνη. Δεν χρειάζεται παρουσία του δράστη, παρουσία του θύματο. Στι κάτω χώρε Έχουμε ένα προηγούμενο που λέγεται υπόθεση Ελχοζούς, όπου ένα Παλαιστίνιο θύμα του, του καθεστώτος Καντάφη ε, πήρε αποζημίωση ενό εκατομμυρίου ευρώ από ένα Ολλανδικό δικαστήριο. Χρειάζεται βέβαια κάποια και οικονομική υποστήριξη από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τώρα, η πρόκληση είναι πώς θα τεθεί σε εφαρμογή, πώς θα εκτελεστεί αυτή η απόφαση. Δεν έχουν συλλεχθεί τα χρήματα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι η διεθνής κοινότητα στέλνει ένα μήνυμα δέσμευσης Υπάρχουν προηγούμενα σε ό,τι αφορά αγωγή αποζημίωση για ηθική βλάβη στι Ηνωμένε Πολιτείε, Καράτζιτ και είχαμε θύματα βιασμού κατά του Ράντεβαν Κάραζιτ ε, και δόθηκαν αποζημιώσεις 740 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν καταβλήθηκαν φυσικά τα χρήματα, όπως ε, καταλαβαίνετε, αλλά δείχνει ότι δίνουμε σημασία σε αυτά τα εγκλήματα. Να περάσουμε τώρα στις διοικητικές κυρώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις, ιδίως κατά τρομοκρατών, ε, έχουν υπάρξει τουλάχιστον από το 1999 κυρώσεις κατά της Αλκάιντα και αφορούν απαγόρευση ταξιδίου δεν μπορούν οι άνθρωποι πια να έχουν διαβατήριο και επίσης μπορεί να δεσμευτούν και τα προσωπικά τους στοιχεία. Ε, αυτές οι κυρώσεις έχουν επιβληθεί και πρόσφατα κατά υποστηρικτών του ISIS. Έχουμε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 2015 σχετικά με το θέμα και φέτος το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα κανονισμό και ο ίδιος ο κανονισμός αναφέρεται στη σεξουαλική βία και αναφέρεται στο βιασμό, στην απαγωγή της σεξουαλική βία, τον εξαναγκαστικό γάμο και την υποδούλωση ανθρώπων. Πιστεύω τώρα η πρόκληση είναι να έχουμε και να αναφέρονται άνθρωποι που αναφέρονται σε αυτή την σεξουαλική βία και όχι απλώς να μιλάμε για τρομοκρατία θα μπορούσε να καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΕΕ να κάνουν περισσότερα και ίσως υπάρχει και μια δυνατότητα να θεωρήσουμε υπεύθυνα τα κράτη. Βέβαια το ISIS δεν είναι κράτος, όμως μπορεί να υπάρχουν κάποια κράτη, δεν θα αναφέρω ονόματα εδώ, που υποβοηθούν το ISIS, το τροφοδοτούν με, εγκλή, με, με όπλα, με συγχωρείτε, και άλλους σπόρους. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνα και αυτά τα κράτη και επίσης ε, κράτη τα οποία απλώς παρακολουθούν και δεν κάνουν τίποτα θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνα. Συρία και το Ιράκ ε, ε, δεν έχουν κάνει ίσως όσα πρέπει για να ελευθερώσουν τις γυναίκες για ζήτη από το ISIS. Έτσι λοιπόν και αυτά τα δύο κράτη θα μπορούσαν να ποινικοποιηθούν επειδή δεν έχουν ασκήσει την επιρροή τους. Τώρα το πλεονέκτημα αυτό είναι ότι έχουν πιο βαθιές τσέπε στα κράτη, όμως ίσω να μην υπάρχει δικαστήριο για να δικάσει ένα κράτο εκτός αν ε, απορρίψει την ε, ασυλία του κράτους. Στον χώρο δικαστήριο είχαμε, παραδείγματο χάρη, μία περίπτωση στο Αμερικανικό Δικαστήριο ε, για την υπόθεση ενό δημοσιογράφου που σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε από το ISIS και ε, ουσιαστικά στην προσφυγή ισχυρίζονται ότι υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ Συρίας και ISIS. Βέβαια δεν έχουμε αυτή τη νομοθεσία στην Ευρώπη και δεν ξέρω αν θα χρειαζόμασταν τέτοια νομοθεσία γιατί είναι κάπως αμφισβητήσιμη η διεθνής νομιμότητα αυτού. Και τέλος, συστάσεις. Η παγκόσμια δικαιοδοσία μπορεί να ενδυναμηθεί, οι μεταναστευτικές αρχές και θα μπορούσαν να συνεργαστούν καλύτερα με τους εισαγγελείς και θα μπορούσαμε να έχουμε πιο συγκεκριμένες κυρώσεις που είναι επικεντρώνουν τη σεξουαλική βία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Τώρα με την άδεια του συμπρόεδρου μου. Ελπίζω θα μιλήσω εκ μέρους των μελών που είναι παρόντα. Πριν σας δώσω το λόγο. Και θα ήθελα να ρωτήσω τους προσκεκλημένους από την μειονότητα των Γεζίντι εάν θέλουν να απευθύνουν ένα σύντομο μήνυμα προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εγώ... Ε, εγώ θεώρησα ότι θα είναι μια γυναίκα. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε Εξ ονόματος αντιπροσωπεία των Γεζίδη, θα ήθελα να σε ευχαριστώ πολύ που μας δώσετε τη δυνατότητα να συμμετάσχω εδώ. Λέγομαι Γεζαντινάη και ασχολούμαι με το θέμα των ε, γυναικών ε, Γεζίδη. Ε, είμαι μέλος της οργάνωσης Airbridge στο Ιράκ και ήρθα χθες κατόπιν προσκλήσεως εδώ και μεταξύ των γεζίδι έχουμε έξι θύματα του ISIS, ορισμένα από εδώ, ε, ορισμένα κάθονται δίπλα μου, πέντε θαραλές νέες γυναίκες οι οποίες ε, κρατήθηκαν από το ίσις μεταξύ τριών και είκοσι μηνών. Ε, το τελευταίο θέμα, ε, κάθε εδώ πλάι μου η, κρατήθηκε από τους γεζίδες οι γονείς της θανατώθηκαν τα αδέλφια της, το, ο μικρός της αδελφός ε, σύρθηκε σε διάφορα στρατόπεδα του ΆΙΣΙΣ, υπευλήθηκαν σε πλήση εγκεφάλου και η Λάμη, όπως σας είπα, ε, κρατήθηκε επί 20 μήνες από το ΆΙΣΙΣ Δυστυχώς ήταν σε ένα ναρκοπέδιο στα σύνορα μεταξύ ε, ε, Κουρδιστάν και περιοχής ελεγχόμενης από το ISIS έχασε το ένα της ε, μάτι, το ένα μεγάλο τμήμα του προσώπου της κάηκε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καθηγητά για την τελευταία σας ε, παρουσίαση, γιατί το Ιράκ και η Συρία είναι υπεύθυνα για τα όσα συνέβασαν. Τώρα έχουμε πάνω από 3.000 γυναίκες και παιδιά που κρατούνται από τον ISIS. Ε, ε, και αν δείτε τι γίνεται στο νόμο, τι προβλέπει ο νόμος στο Ιράκ, δεν θα βρείτε κανένας, καμία διάταξη του νόμου που να έχει σαν σκοπό να τιμωρηθούν οι δράστες. Εγώ είμαι φυσικός επιστήμων, δεν είμαι νομικός, αλλά ε, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν ε, να καταδικαστούν για βιασμό μόνο σε έξι, για έξι μήνες και σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο μπορούν να διαφύγουν αυτή την ε, ποινή. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ούτως ώστε να υπάρξει κάποια ποινική λογοδοσία για τέτοια εγκλήματα κατά τον Γεζίντι. Τα κορίτσια αυτά που βρίσκονται εδώ θέτουν συνεχώς το ερώτημα πότε θα έρθει η ώρα να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Και θεωρώ ότι είναι και ευθύνη της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά να κάνει μια συγκεκριμένη έκκληση ε, για αυτά τα κορίτσια. Υπάρχει ένα κορίτσι 9 ή 10 ετών που όχι μόνο βιάστηκε αλλά έμεινε έγκυος από μαχητή του Άισις. Εγώ έρχομαι από μια αγροτική κοινότητα, είναι πολύ απλοί άνθρωποι, ε, ζούσαμε σε πολύ ειρηνικές συνθήκες εδώ και 5.000 χρόνια και τώρα οι άντρες μας ε, θανατώθηκαν. Ένας ε, ο οποίος επέζησε ήταν αυτόπτης μάρτυρας το, της θανάτωσης όλων των αντρών. 400 άνδρες ήταν ε, και αυτός ήταν ο μόνος επιζήσας. Η Λάμια είναι ανιψιά του, αυτός έχασε όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Τώρα, το ερώτημα προς τη διεθνή κοινότητα είναι το εξής. Εάν περιμένετε το Ιράκ να ε, τυθεί να ε, γίνει μέλος, αυτό δεν προτίθεται να το κάνει το Ιράκ. Το Ισλάμ είναι κατά του να υπάρξει ποινή, να, να καταδικαστούν τα μέλη του ISIS. Πέρσι είχαμε πάνω από 3.000 τέτοιες γυναίκες και παιδιά και ήταν σε απόσταση μόνο 7 χιλιόμετρα από τις ε, κουρδικές δυνάμεις και τις δυνάμεις των συμμάχων και κανείς απολύτως δεν προσπάθησε να διανύσει αυτή την απόσταση για να απελευθερώσει αυτές τις γυναίκες και τα παιδιά. Εάν... Γιατί οι γυναίκες αυτοί, αυτές και τα παιδιά ε, μεταφέρονται σε άλλες περιοχές που ελέγχονται πλήρως από το ISIS, όπως τη Ράκα κλπ. Τώρα, ε, άρχισαν τέτοιου είδου επιχειρήσει απελευθέρωσης αυτών των γυναικών, αλλά είναι ελάχιστες αυτές οι οποίες απελευθερώθηκαν ίσω μία ή δύο τέτοιες περιπτώσεις. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω ότι αυτή η ακρόαση ε, θα σας δώσει κάποια ελπίδα ότι προσπαθούμε να βρούμε νόμιμους τρόπους, τα ένομα μέσα, ούτως ώστε να τιμωρηθούν αυτά τα εγκλήματα. Παρόλο στη νομική στεκή γλώσσα είναι δύσκολο είναι δύσκολο να παρακολουθεί αυτή η νομική γλώσσα. Έχω την κυρία Χάουταλ εδώ, η οποία ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς το πώς ε, προσλαμβάνουμε τα όσα μας είπατε και την παρουσία σας εδώ. Παρ' όλα αυτά, ε, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πολύ θετικά σημεία. Η Νάντια Μούρατ ήταν μία από τις ε, υποψήφιες, μία από τις υποψήφιες για το βραβείο Ζαχάροφ και επίσης ε, ε, ελήφθη η πρωτοβουλία να σταθεί μια ομάδα φιλίας με τους Γιαζίντι. Θα ήθελα να, ερωτη... να απευθύνω κάποια ερωτήματα προς τους τρεις νομικούς εμπειρογνώμων τους οποίους ακούσαμε. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν σε θέση να, να θαρρύνει και να παρατηρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει δράση Ποια θα ήταν τα στοιχεία κλειδιά που εμείς ως Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να κάνουμε, ούτε ώστε να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να κάνει αυτό το οποίο υποχρεώται να κάνει υπό το διεθνές δίκαιο, ούτως ώστε να θέσει ένα τέρμα στην ατιμερουσία και τις οδύνες αυτών των ανθρώπων. Ε, αναφέρθηκε ότι υπάρχει μια παγκόσμια δικαιοδοσία, αλλά θα πρέπει, η, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι δράστες θα πρέπει να είναι παρόντες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ μεταναστευτικών και δικαστικών αρχών. Εμείς έχουμε τη Eurojust, η οποία ερευνά τέτοιου είδου διασυνορικές υποθέσεις. Είναι κάτι το οποίο εσείς θα θέλετε να ενθαρρύνετε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης. Το ερώτημά μου είναι επίσης πάνω από 100 βουλευτές έγραψαν προς τη Φρεντερίκα Μοργκερίνη ζητώντας της εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ορίσει τα εγκλήματα κατά τον γεζίδη, ειδικά ε, να τα χαρακτηρίσει, ειδικά τα εγκλήματα κατά γυναικών και παιδιών, σαν ε, μορφή γενοκτονίας. Ε, και πολλά όργανα των Ηνωμένων Εθνών ε, χώρες μέλη και τρεις τρίτες χώρες το ζήτησαν. Αλλά η κυρία Μοργκερίν δεν ε, απάντησε στην επιστολή αυτή την οποία στείλαμε τον Απρίλιο. Ε, και πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την συνεργασία με το Τμήμα Δικαιοσύνης γιατί πραγματικά θα πρέπει να, υπάρξουν, να υπάρξει ανάληψη ευθύνη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ο Συμπρόεδρος έχει να κάνει μια ερώτηση. Δύο ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Προς τους ομιλητές. Καταρχήν βέβαια θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Σε ό,τι αφορά αυτές τις μαρτυρίες τις οποίες ακούσαμε και στα θύματα διώξεων. Και σφαγών, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν και γενοκτονία. μία ερώτηση ό,τι αφορά την νομιμοποίηση, την αξιοπιστία και την ικανότητα των διεθνών ποινικών δικαστηρίων. Πώς ε, αξιολογείται αυτή η αξιοπιστία, η νομοποίησή τους υπό το φως της, ε, του γεγονότος ότι 20 χρόνια μετά το τέλος της σύγκρουσης στην πρώην Ιγκοσλαβία, της, ε, και 10 χρόνια μετά το θάνατό του της αθώσεις του Μιλόσεβιτς που έγινε τον Αύγουστο από, για εγκλήματα στην πρώην Οικοσλαβία Ε, αυτό αποτελεί αποτέλεσμα ε, εξωτερικών παρεμβάσεων. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το γεγονός, για αυτό το επεισόδιο. Άλλη ερώτηση. Από ό,τι φαίνεται και οι τρεις ομιλητές αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που υπάρχουν ε, να δώσουμε έναν νομικό ορισμό ε, των προτεργατών και των θητών γενικά, γενικότερα. με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό και πώς μπορεί να βοηθήσει το διεθνές δίκαιο, πώς μπορούν να βοηθήσουν πώς μπορεί να βοηθήσει το διεθνές δίκαιο ε, σε ό,τι αφορά την μεταχείριση των κρατών που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν αυτές τις δράσεις. Η διεθνή κοινότητα, για παράδειγμα, σήμερα μπορεί να αναγνωρίσει ε, την ε, ευθύνη της Σοβιετικής Ένωσης για τη δημιουργία των Ταλιμπάν πριν από 40 χρόνια. Μετά, ο κ. Ζενγκάρ, δεν είμαι σίγουρος αν ε, προφέρω σωστά το όνομά του, ε, ο κ. Ριγκάρτ, ε, ε, αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική κρίση. Εγώ δεν μίλησα. Δεν συνέδεσα αυτή την κρίση με τη ριζοσπαστικοποίηση και την ε, τρομοκρατία. Όμως είπε ο κ. Ζενγκάρτ ότι ορισμένοι από αυτούς τους εγκληματίες φτάνουν στην Ευρώπη μέσω μεταναστευτικών ροών. Υπάρχουν αποδείξεις έστω και μία απόδειξη για κάτι τέτοιο. Εμείς δεν γνωρίζουμε κάποιο τέτοιο στοιχείο. Εγώ θα έλεγα, αντιθέτως, ότι οι τρομοκράτες οι, οποίες, οι οποίοι προέβησαν σε τρομοκρατικές πράξεις σε ευρωπαϊκό έδαφος, σίγουρα δεν πέρασαν, δεν διέσχισαν τη Μεσόγειο με σκάφη, ε, όπως ε, πολλοί άλλοι πρόσφυγες. Έφτασαν μάλλον με άλλο τρόπο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. κυρία Ντελβό, ε, είναι δύσκολα τα λόγια μετά από αυτές τις ε, μαρτυρίες, συγκινητικές μαρτυρίες που ακούσαμε. Ε, πώς να παρηγορήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να προλάβουμε τέτοιου είδου εγκλήματα στο μέλλον. Γιατί οι διώξεις και η τιμωρία δεδομένης και της καθυστέρησης δικαιοσύνης πιστεύω ότι δεν είναι αρκετές. Και θα είναι και καθυστερημένες. Αυτό όμω δεν αποτελεί λόγο για να αποφύγουμε την εμπλοκή μας. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τιμωρήσουμε ε, και να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Καταλαβαίνω ότι οι διεθνείς διαδικασίες είναι πολύ αργές και τους επόμενους, αλλά τους επόμενους μήνες χρειάζεται να προσπαθήσουμε να αποδοθεί διεθνής δικαιοσύνη. Ήθελα όμως να σχολιάσω αυτό που ο κ. Ρίγκαρτ έδωσε παραδείγματα συνεργασίας ανάμεσα σε υπηρεσίες μετανάστευσης και ε, τη δικαιοσύνη και ανέφερε τις κάτω και τη Γερμανία πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα να ρωτήσω, Τέτοιου είδους συνεργασία υφίσταται και σε άλλα κράτη-μέλη. Και σε ποια βάση γίνεται αυτή η συνεργασία. Ε, πρόκειται για την τιμωρία ε, ε, αδικημάτων που έχουν διαπραχθεί στην ίδια χώρα και τώρα ή και στο παρελθόν. Πρόεδρος. Θα ήθελα οι ομιλητές να είναι συντομοί και συνοπτικοί γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ίσως θα ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση, τη συνεργασία μεταξύ μεταναστευτικών αρχών και διοκτικών αρχών. Εγώ ανέφερα το Ολλανδικό και το Γερμανικό παράδειγμα γιατί είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Σίγουρα υπάρχουν και σε άλλα μέρη, αλλά θα πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά. Αλλά βασίζονται στο άρθρο 1F που λένε ότι κανείς δεν μπορεί να έχει καθεστώς ε, πρόσφυγας εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει εμπλακεί σε εγκλήματα. Ε, και πολύ συχνά ε, οι άνθρωποι αυτοί διώκονται ε, και ε, ενώ αυτοί έχουν διαπράξει κάποιες ε, πράξεις αλλού, ενώ εδώ θα πρέπει να επικεντρώσουμε σε πράξεις που έγιναν στη Συρία και στο Ιράκ. Κύριε Συμπρόεδρε, νομίζω ότι έγινε μια παραξήγηση. Ενδεχομένως υπάρχουν δράστες που κάνουν σεξουαλικά εγκλήματα τα οποία περνούν μέσω των ροών των προσφύγων. Ε, βεβαίως ε, υπάρχουν ε, εγκληματικές συμμορίες οι οποίες ε, διοχετεύουν αυτές τις προσφυγικές ροές. Τώρα, τι μπορούν να κάνουν οι εμπειρογνώμονες. Σας έδειξα την τελευταία διαβάνα και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε πολλές φορές ότι θα πρέπει να συσφιχθεί η συνεργασία στις χώρες μέλη μεταξύ διοκτικών και μεταναστευτικών αρχών. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να στηρίξει τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Γιατί πολύ συχνά ε, εξαρτώνται ακόμα και αρχές από την υποστήριξη των ΜΚΟ. ε, πολλές φορές ε, έγινε μνήα για νέο απικιακά σχήματα. Αλλά εγώ θα πρέπει να το αρνηθώ. Είδαμε τι έγινε με το δικαστήριο της Χάκης, πόσο πολύ άργησε. Ίσως θα πρέπει να αναμένουμε μέχρι το τέλος της σύγκρουσης, ούτω ώστε να συσταθούν τέτοιου είδου θεσμικά όργανα και θα πρέπει να υπάρχει δικαιοδοσία στο επίπεδο των χωρών μελών. Επίσης, ε, θα πρέπει όσον αφορά τις κυρώσεις έναντι εκείνων που υποστηρίζουν τη δημοκρατία, εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλοι κατάλογοι, αλλά δεν πρόκειται για μια γενική σχέση υποστήριξη ή ίσως οικονομική υποστήριξη προς τους τρομοκράτε, αλλά θα πρέπει, εφόσον αυτή συνδέεται με την διάπραξη σεξουαλικών εγκλημάτων. Θα ήθελα να το θέσω στο εξή πλαίσιο, να πω. Καμιά από αυτές τις ε, προκλήσεις Θα ήθελα να ξεκινήσω και πάλι. Όσον αφορά το ζήτημα της παγκόσμιας δικαιοδοσία. Αυτό συνέβη σε σχέση με πολλές άλλες ε, έναπλες ε, συγκρούσεις. Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές ε, συνήθως δεν διώκονται αποτελεσματικά, ιδιαίτερα όσον αφορά με περιπτώσεις άσκησης σεξουαλικής βίας. Και υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις στη Γερμανία είναι πολύ δύσκολες ε, περιπτώσεις να διωχθούν στο πλαίσιο των εθνικών δικαιοδοτικών οργάνων, όχι μόνο λόγω των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά και της έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης, το θέμα του, του βαθμού του δικαστηρίου, της ε, παρκούς ε, δικαιοδοτικής αρμοδιότητας κλπ. Αυτό δεν είναι επιχείρημα για να μην διωχθούν αυτές οι περιπτώσεις, αλλά σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους. Το δεύτερο το, της δίωξης, το δεύτερο που θα ήθελα πω είναι το εξή. Πράγματι, το δικαστήριο της πρώην Ιουκοσλαβίας συστάθηκε κατά τη διάρκεια της ε, σύγκρουσης. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει να ακολουθήσει ένα αντίστοιχο δρόμο, ίσως η ενδεδειγμένη χρονική στιγμή θα ήταν τώρα και μάλιστα σε σχέση με την άσκηση πίεση εκ μέρους της ε, διεθνής ε, ε, κοινότητας. Αυτά είναι διεθνή εγκλήματα και εγώ θα χαρακτήρισα εγκλήματα σεξουαλικής βίας οι εγκλήματα στη βάση του φύλου να τα ξισώσω με τα τρομοκρατικά εγκλήματα το διεθνές ποινικό δίκαιο δεν εξετάζει μόνο τη ριζοσπαστικοποίηση, και την ε, τρομοκρατία ε, σε σχέση με αυτά τα εγκλήματα, αλλά ε, και την άσκηση βίας αυτή καθ' αυτή. Προφανώς ε, δεν μπορούμε να ε, ε, εκφράσουμε εμεί, να αποφαθούμε για την οδύνη των θυμάτων. Όσον αφορά την αξιοπιστία των διεθνών δικαστηρίων, η διεθνής δικαιοσύνη δεν είναι αποτελεσματική, οι διώξει θα πρέπει να βελτιωθούν. Για παράδειγμα, το δικαστήριο της πρώην Ιγκοσλαβίας και το δικαστήριο για τη Ρουάντα, εκεί ήταν πολύ χρονοβόρες οι διαδικασίες. Ε, πάντοτε ήταν πολύ χρονοβόρες σε εθνικό επίπεδο. Ε, σε χρονικό επίπεδο οι διαδικασίε είναι πολύ πιο σύντομε. Άρα θα πρέπει να ενισχυθούν οι διαδικασίε αυτέ, οι ποινικέ διώξει. Θα πρέπει οι χώρε να κινητοποιηθούν, ούτε ώστε οι διώξει αυτέ, οι δίκε αυτέ να συντομευθούν. Δεν είναι δυνατόν να διαρκούν τρία ή τέσσερα χρόνια και η δικαιοσύνη χάνει την αξιοπιστία τη. Τώρα, όσον αφορά την νομιμότητα, αυτό είναι πολύ σύνθετο θέμα. Και ε, θεωρώ ότι εδώ έχουμε μια πολύ φιλόδοξο, ένα πολύ φιλόδοξο όραμα, φιλόδοξη ιδέα εν σχέση με τη ε, διεθνή δικαιοσύνη. Η διεθνή δικαιοσύνη ε, θα πρέπει να περιοριστεί να επιτελεί το έργο της, δηλαδή να απονέμει δικαιοσύνη. Ε, και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί και η υπόλοιψή της. Ωστόσο, όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, κανείς δεν πίστευε ότι οι υπεύθυνοι τελικά θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα, ε, βεβαίως υπάρχουν ε, Υπάρχει μια εξέλιξη στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στο Λίβανο. Πρόσωπα τα οποία ε, συμμετείχαν εκεί ε, στον πόλεμο συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών. Άρα εκεί δεν έχει υπάρξει τέτοιου είδους ε, κοινωνική εξέλιξη. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους δικαιοδοτικά όργανα, αλλά των οποίων η αξιοπιστία θα πρέπει σίγουρα να ενισχυθεί. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία σας. Οι συζήτησεις αυτές ήταν πολύ χρήσιμες, νομίζω, για μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την αντιπροσωπεία των Γιαζίδης. Ελπίζω ότι φεύγετε τουλάχιστον με την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό σας και ότι προσπαθεί να διώξει και να τιμωρήσει ε, τα δικήματα που δεν πράχθησαν εις βάρος σας. Ευχαριστώ πολύ.